Ruhig, I think we can start. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe meine sehr geehrten Damen und Liebe συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής ΤΡΑΝ. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Έγκριση των πρακτικών της 1ης Σεπτεμβρίου. Και εδώ πέρα, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται τα πρακτικά. Για τις ανακοινώσεις από την συνεδρίαση των συντονιστών ε, της 1ης Σεπτεμβρίου έχετε λάβει αντίγραφα. Αν δεν έχετε μέχρι τις 5.30 ώρα κάποια αντίρρηση, εγκρίνονται και αυτά. Μετά, να πω πως την 5η, 11 η ώρα, θα έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή των Περιφερειών για διασυνοριακές συνδέσεις που λείπουν συγκοινωνιακές συνδέσεις. Ξέρετε ότι είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, έχουμε ασκήσει πίεση και στην Κομισιόν και η Κομισιόν έχει κάνει μια πρόταση και θέλει να διαθέσει 110 εκατομμύρια ευρώ και η Επιτροπή των Περιφερειών πάντα μας στήριζε εδώ. Γι' αυτό έχουμε μια κοινή συνεδρίαση και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κάθε έναν από εσά να είστε εδώ πέρα την ε, Πέμπτη παρόντες γιατί βεβαίως δεν είναι ωραίο να είμαστε δύο-τρεις μόνο. Πέμπτη 11 η ώρα λοιπόν. Σας παρακαλώ κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή των Περιφερειών. Περνάμε τώρα στο σημείο 4. Δύο θέματα Στατιστικά για τις μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών και στατιστικά σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές όσον αφορά την συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα επιβάτες και ατυχήματα. Εδώ πέρα πρέπει, σύμφωνα με τον κανονισμό, να πω κάποια πράγματα για διαδικασία. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου στις 15 Σεπτεμβρίου Ε, γνωστοποίησε την ε, συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 66.2 προβλέπονται τα εξής. Η θέση του Συμβουλίου θα μπει ως πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης της Αρμόδιας Επιτροπής μετά, που θα συνεδριάσει μετά από την γνωστοποίηση. Εδώ έχουμε λοιπόν σήμερα την πρώτη συνεδρίαση και το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι αυτό. Οπότε, σας ανακοινώνω επίσης σήμερα πως ε, μας έφτασε η θέση του Συμβουλίου και άρα ξεκινάει η δεύτερη ανάγνωση για αυτή την νομοθετική ε, πρόταση. Και η ψηφοφορία θα λάβει χώρο στις 11 ε, Οκτωβρίου. Συμφωνείτε όλοι. Ωραία, περνάμε τώρα σημείο 5 η βελτίωση των συνδέσεων και της προσβασιμότητας των μεταφορικών υποδομών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Έκθεση πρωτοβουλία, πρωτοβουλίας, ο κύριος Πορέμπα. Περνάμε στην ψηφοφορία, η οποία πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε τα μηχανήματα. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Ωραία. Σα. ευχαριστώ. Λοιπόν, συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 18 ναι, υπέρ, 12 κατά, Δύο εποχές, συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέγγι 13 μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ρέγγι 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ε, τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να την απολυτεύσουμε. 63. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 12 υπέρ, 20 κατά, απορρίπτεται. Αλλά ε, σας παρακαλέσω τότε να σηκώνετε ψηλά τα χέρια. Ρέγγι 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 65 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ρέγγι 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή ρέγγι 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή ρέγγι 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή ρέγγι 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή ρέγγι 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές να την επαληθεύσουμε. 73 Άρχιτε η ψηφοφορία. Πέρας. 19 υπέρ, 12 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβασική 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε 95 άρχεται Πέρας. 12 υπέρ, 20 κατά, καμία αποχή απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. εποχές Δεκτή. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ορίστε. 99 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 18 υπέρ, 15 κατά καμία αποχή δεκτή. 100 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 102 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 120 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 23 επερ Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 96 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 24 υπέρ. Κατά εποχές δεκτή. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά εποχές δεκτή. 133 υπέρ. Κατά εποχές δεκτή. 134 υπέρ. Κατά εποχές δεκτή. 135 υπέρ. Κατά εποχές δεκτή. 136 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα συμβαστική 26. Εδώ πέρα μου έχει πει ο εισηγητής ότι στην συνεδρίαση των σκιωδών δεν υπήρξε κοινή θέση για το εάν θα γίνει θα μπει στη συμβαστική πρόταση το κομμάτι για τον θόρυβο. Γι' αυτό θα ψηφίσουμε αν θα μπει στη συμβαστική πρόταση αυτό το κομμάτι η περίοδος που αφορά τον θόρυβο. Υπό παραγραφός 17 και να λάβει τα μέτρα για την ανάπτυξη του ERTMS καθώς και για τη μείωση του θορύβου στις εμπορευματικές μεταφορές. Ποιος είναι υπέρ του να μπει αυτή η μη περίοδος. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι, όχι, πρώτα αυτή την περίοδο. Πέρας. 13 υπέρ, 18 κατά, δύο αποχές. Απορρίπτεται. Και άρα ψηφίζουμε την συμβαστική 26 ε, χωρίς αυτή την προσθήκη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 147 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. 147. Άρχεται. Πέρας. 11 υπέρ, 20 κατά, 2 αποχές. Απορρίπτεται. Ε, συμβαστική 27 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 156 υπέρ. Κατά. Άποχες. Να την επαληθεύσουμε. 156. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 11 υπέρ, 9 κατά, 13 αποχές δεκτή. Συμβαστική 29 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 160 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ρέγγι 10 μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή 163 υπέρ κατά αποχές δεκτή 165 υπέρ κατά αποχές δεκτή 166 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβασική 30 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 31 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 32 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. 186. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ, 10 κατά, 3 άποχες, εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά, άποχες, και αυτό θα το επαληθεύσουμε 185 άρχεται η ισοφορία πέρας 22 υπέρ 10 κατά μία αποχή εγκρίνεται συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε και αυτήν άρχεται η ψηφοφορία για την 192 πέρας 22 υπέρ 11 κατά καμία αποχή εγκρίνεται συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. Ρέτζι 11 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την απολυτεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία από τις 18. Πέρασε. 19 υπέρ, 11 κατά, 2 εποχές συγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά, αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. 28 υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Πορέμπα. Θα προχωρήσουμε τώρα στην ανταλλαγή απόψεων. για το θέμα του κ. Σκέλετς, τον οποίο δίνω τον λόγο. Πρόκειται για την προσέγγιση νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων κρατών μελών όσον αφορά τι απαιτήσει προσβασιμότητα για τα προϊόντα και τι υπηρεσίε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ορίστε, ορίστε κύριε Σκέρλες. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να επενέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο της προτείνει, ε, δηλαδή υποβάλλει μια πρόταση οδηγία, υψηλή ποιότητα ποιότητας για την προσέγγιση των νομοθετικών και άλλων διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά απαιτήσει προσβασιμότητα για προϊόντα και υπηρεσίε, και ω συζητητής θεωρώ ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η υποδομή ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και σε μεταφορές και ε, τουρισμό για όλους τους ανθρώπους που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην διακήρυξη των Ενωμένων Εθνών για τα δικαιώματα ανθρώπων με αναπηρίες προτείνονται και κανόνες. Και εμείς πιστεύουμε σε αυτό και αναμένουμε ταχεία ψήφιση των διατάξεων για την προσβασιμότητα. Η οδηγία αναφέρεται και στην προσβασιμότητα από πλευρά προσώπων με αναπηρίες ή με λειτουργικές αδυναμίες σε ζητήματα μεταφορών και τουρισμού. Πρέπει να επιμείνουμε στις, ε, στην ανάγκη προσβασιμότητας και όταν περνούν οι άνθρωποι αυτοί από, μια, από ένα τρόπο μεταφοράς σε άλλο, πρέπει και εκεί να είναι δεδομένη η προσβασιμότητα, καθώς επίσης και σε, στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδες για να μπορέσουν να αγοράσουν εισιτήρια, και ούτω καθεξής. Δηλαδή προσβασιμότητα και σε όλες τις σύγχρονες υπηρεσίες προσφέρει το διαδίκτυο και άρα και διασυνδεσιμότητα. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε διακρίσεις. Θα επιτευχθεί δε αυτό μόνο εφόσον υπάρχει προσβασιμότητα στις υποδομές ε, του, του τουρισμού και στις πολυτροπικές μεταφορές. Η προσβασιμότητα είναι πολύ σημαντική για τον τομέα του τουρισμού, για να μπορέσει ο κάθε άνθρωπος να έχει πρόσβαση και στις υπηρεσίες που προσφέρει ο τουρισμός. Είμαι λοιπόν βέβαιος ότι σε συνεργασία με τους κοιόδης συγητές θα επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα στην σύνταξη της νομοδοτήσεως της παρούσης Επιτροπής, κάτι που πιστεύουμε ότι θα ε, βελτιώσει και την προσπάθειά μας στον αγώνα κατά των διακρίσεων σε βάρος των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ και αναμένω τη συνεργασία με τους κοιόδης συγητές. Τώρα βέβαια πριν να δώσω το λόγο στους κοιόδης ζήτησε τον λόγο η εκπρόσωπος της ε, Κομισιόν, κυρία Πορέρο. Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε συντόμως το νομοθέτημα για την προσβασιμότητα. Έχουμε επισκεφθεί και άλλες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές, την Επιτροπή Προστασία Καταναλωτών και του Περιβάλλοντος και επειδή είναι σημαντική η προσβασιμότητα και για τις μεταφορές, για αυτό βρισκόμαστε και σήμερα εδώ. Στα πλαίσια της στρατηγικής για την διευκόλυνση των αναπήρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε πρωτοβουλία για να βελτιώσει τις υποδομές και μεταξύ των οκτώ προτεραιοτήτων της στρατηγικής οι υποδομέ είναι η πρώτη. Η στρατηγική προβλέπει ότι η Επιτροπή θα διερευνήσει τις δυνατότητες λήψεως ρυθμιστικών μέτρων για την επιβολή ειδικών προδιαγραφών για τους διάφορους τομείς, ώστε να διευκολυνθεί και η προσβασιμότητα, γιατί αυτό υπαγορεύει και η νέα αγορά. Η βελτίωση της ενιαίας αγοράς θα έχει και θετικές επιπτώσεις στην διευκόλυνση και το έργο της βιομηχανίας, αλλά πρωτίστως θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ισότητα, στην ίση μεταχείριση προσώπων με αναπηρίες, διότι πρόκειται για 18 εκατομμύρια ανθρώπους, περίπου το 20% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Όλες οι χώρες μέλη, εκτός μιας η οποία ολοκληρώνει τώρα την διαδικασία, έχουν κυρώσει την Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τη διευκόλυνση των ε, αναπήρων και αυτή η συμφωνία επιβάλλει και την βελτίωση των υποδομών για προσβασιμότητα και με συγκεκριμένα πρότυπα προδιαγραφές καθώς και με συγκεκριμένες προθεσμίες για την παρακολούθηση, το monitoring δηλαδή. Για να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις αυτές χρειάζονται κοινοί κανόνες στο ευρωπαϊκό επίπεδο διότι αυτό θα βοηθήσει να αποφευθούν αποκλήσεις στην ομοθεσία και κατακαιρματισμός της ενίας αγοράς. Αυτοί που θα εποφεληθούν πρωτίστως είναι η βιομηχανία και οι κατασκευαστές και αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες, διότι με κοινά πρότυπα, κοινές προδιαγραφές θα διευκολυνθεί το έργο τους και θα έχουν και ασφάλεια δικαίου, ότι δηλαδή τα προϊόντα τους εκπληρούν τις ε, ε, διατάξεις και προδιαγραφές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλοι που θα ε, ωφεληθούν θα είναι βεβαίως οι ίδιοι ανάπηροι καθώς και ηλικιωμένοι. Ας μην λησμονήσουμε ότι και οι χώρες μέλη με ειδικέ λύσεις, ειδικέ λύσεις, εξειδικευμένες λύσεις δηλαδή, είναι πιο δαπανηρές. Γι' αυτό εάν συμφωνήσουν με την προσπάθεια που κάνουμε να δοθούν λύσεις για όλους, θα διευκολυνθούν και θα έχουν και μικρότερο κόστος. Μια, για παράδειγμα, ένας αυτόματος πολιτής εισιτηρίων που είναι ευκολότερα προσβάσιμος, διευκολύνει όλο τον κόσμο. Ή, για παράδειγμα, το να μπορεί κανείς να αντλήσει πληροφορίες από ένα μηχάνημα σε ένα θορυβόδες ε, περιβάλλον, σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό. Εφόσον διευκολυνθεί εκεί, αυτό διευκολύνει όλους μας. Από τη βιομηχανία θα υποφεληθούν περισσότερο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι με ένα ενιαίο σύνολο κανόνων θα τις βοηθήσουμε ώστε να συμμετέχουν και σε διαμεθοριακές ενέργειες. Θα χρειαστεί λοιπόν ε, ε, να δαπανούν και λιγότερο για να προσαρμόζονται στις διαφορετικές νομοθεσίες των διαφόρων χωρών μελών. Το νομοθέτημά μας έχει δύο σκέλη. Το πρώτο επιβάλλει υποχρεώσει προσβασιμότητας σε ένα αριθμό προϊόντων και υπηρεσιών και επιβαρύνει τους επιχειρηματίες, τη βιομηχανία και ούτω καθεξής. Το δεύτερο σκέλος χρησιμοποιεί τις ίδιες απαιτήσει προσβασιμότητας που είναι λειτουργικές και διευκρινίζει την έννοια της προσβασιμότητας σε όλο το ευρωπαϊκό δικαιικό οικοδόμημα, για παράδειγμα και για ε, διαδικασίες προμηθειών. Ποια είναι τα βασικότερα στοιχεία του νομοθετήματος όπως είπα, αφενός έχει τις λειτουργικές απαιτήσεις προσβασιμότητας που συνδυάζονται με ρήτρα που διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών που πληρούν αυτές τις προδιαγραφές. Σε ό,τι αφορά με τη συμμόρφωση, πρώτα-πρώτα ξεκινά με την αυτοδιακήρυξη, αυτοδήλωση, ότι δηλαδή ο κατασκευαστής δηλώνει από μόνος του ότι συμμορφούνται και προχωρά σε άλλα στάδια έγκριση και από τις ε, αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ή ε, δυνατότητα υποβολής καταγγελιών από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις αναπήρων προσώπων. Αυτό που δεν κάνει το νομοθέτημά μας είναι δεν μπαίνει στις τεχνικές λεπτομέρειες των λύσεων. Αφήνει τους επιχειρηματίες, τους φορείς που θα ε, λειτουργήσουν υπό τις, υπό τις διατάξεις αυτές να αποφασίσουν ποιες είναι οι σωστές λεπτομέρειες, τεχνικές λεπτομέρειες. Και δεν επιβάλλει επίσης βάρη και απαιτήσει. Δηλαδή περιλαμβάνει διατάξεις για την δυσανάλογη επιβάρυνση. Δεν τροποποιεί, τροποποιεί δε την τομιακή νομοθεσία. Αλλά παρεμβαίνει συμπληρωματικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζει την σύνταξη του νομοθετήματος της, της προτάσεως της, για να το πράξει αυτό δηλαδή εξέταση της νομοθεσίας όρων των χωρών μελών και προέβηκε και σε βάθος μελέτη των χωρών μελών και τους τομείς και, τον, και τους οικονομικούς τομείς που φτάνουν το 80% συνολικά του ευρωπαϊκού ΕΠ και κατέληξε στο ότι υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκό νομοθέτημα όπως η οδηγία. Σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση με τις διατάξεις των δημοσίων προμηθειών, αυτές απαιτούν ήδη να επιβάλλεται η προσβασιμότητα και στις προσκλήσεις εκδόσεις ενδιαφέροντος. Το ίδιο συμβαίνει και στις διατάξεις των διαθωτικών ταμείων και στις περιπτώσεις όπου οι δημόσιες αρχές αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν την προσβασιμότητα για τις δημόσιες μεταφορές. Το Accessibility Act δεν τροποποιεί τον εθελοντικό χαρακτήρα των άλλων αυτών διατάξεων, νομοθετικών διατάξεων. Συνδέεται και με την οδηγία προσβασιμότητας στο διαδίκτυο και επιβάλλει ακριβώς τις ίδιες απαιτήσεις Όπως είπα πριν, περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερο άρθρο για την αναλογικότητα και επικουρικότητα και με την προσεκτική επιλογή των προϊόντων, με την εφαρμογή των απαιτήσεων στα νέα προϊόντα, με την παροχή υπηρεσιών από μια ημερομηνία και μετά, ε, περιλαμβάνει και διατάξεις για τη συμμόρφωση και ούτω καθεξής. Έχω και μια τελευταία διαφάνεια για την εφαρμογή. Λέμε δύο χρόνια μετά από την θέση ισχύ και έξι χρόνια για την εφαρμογή. Και έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας πέντε χρόνια μετά από την έναξή της. Ευχαριστώ πολύ που με επιτρέψατε να σας αναπτύξω με λίγα λόγια τον στόχο της οδηγίας. Ευχαριστώ. Λίμπλιχ Κόχ. Ο κύριος Κόχ δηλαδή. Ευχαριστώ και τον εισηγητή την, και την ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν. Χαίρομαι για την πρωτοβουλία της ε, Κομισιόν που ενισχύει τα δικαιώματα των αναπήρων και την συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την ε, ε, διευκόλυνση των αναπήρων, αυτή ήδη αναφέρθηκε και αυτό είναι σημαντικό και για την προσβασιμότητα και στις διάφορους, στους διάφορους τρόπους μεταφορών. Δύο σύντομες ερωτήσεις λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πρώτη, πώς θα εμποδίσει η Κομισιόν να έρθουν οι νέες αυτές διατάξεις σε αντίθεση με διατάξεις που ισχύουν ήδη για τα δικαιώματα των επιβατών και δεύτερο για το πεδίο εφαρμογή. Πρόσωπα με μείωση της λειτουργικότητάς τους επιλέξει. Ε, ρωτώ, είναι ευρύτερο το πεδίο εφαρμογή από αυτά που έχουμε χρησιμοποιήσει ως τώρα, δηλαδή άνθρωποι με αναπηρίες ή άνθρωποι με περιορισμένη κινητικότητα. Αυτά που απορρέουν δηλαδή από τις διατάξεις που ισχύουν ήδη, για παράδειγμα, για τα δικαιώματα των επιβατών. Δηλαδή, με τη νέα αυτή ε, πρόταση που κάνετε, προσπαθείτε να περιλάβετε και, για παράδειγμα, εγγύους ή ανθρώπους οι οποίοι προσωρινά είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν κάποιο βοήθημα για να βαδίσουν ή κάτι τέτοιο. Αυτό δεν είναι σαφές για μένα. Όργα ανάλογα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση της Επιτροπής στη δική μας Επιτροπή και ευχαριστούμε και τον εισηγητή. Συνεργαστήκαμε στη σύνταξη και προγενέστερων εκθέσεων. Οι μεταφορές ε, είναι ύψης της σημασίας για ανθρώπους με αναπηρίες. Γι' αυτό και η πράξη προσβασιμότητας θα πρέπει να λάβει υπόψη και αυτή την πτυχή. Μιλάμε για προϊόντα και για υπηρεσίες μεταφορών. Δεν μιλάμε μόνο για αμαία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις υποδομές για την προσβασιμότητα σε όλα τα είδη των μεταφορών. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς έχει υπάρχουσα νομοθεσία. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της μεταφορές θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις τεχνολογίες που υποβοηθούν τους ανθρώπους με αναπηρίες, έτσι ώστε να μην υπάρχουν περισσότερα προσκόμματα. Περιμένω την περαιτέρω συνεργασία με τον εισηγητή και τους συναδέλφους, διότι αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ σημαντική για 80 εκατομμύρια ανθρώπους με αναπηρίες, αλλά και για όλους εμάς. Τζάκι Φώστερ. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή. Νομίζω ότι όλοι καλωσορίζουμε αυτά τα μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης πρόσβαση όλων και να μπορούν να ε, μεταβαίνουν όπου επιθυμούν με την ίδια ευκολία και τα άτομα με αναπηρία. Ξέρουμε και συμφωνούμε με το θέμα αρχής, αλλά ως προς τη, την έκθεση της Επιτροπής θα ήθελα να πω ότι δεν καταλαβαίνω τι εννοείται σε πολλές, στη σύνταξη ορισμένων προτάσεων πολλές φορές ε, υπάρχει γλωσσικό θέμα. Όταν χρησιμοποιείται ορισμένους επιθετικούς προσδιορισμούς σε σχέση με δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καταναλωτές και επιβάτες. Επίσης, αυτό το πέρασμα της νομοθεσίας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχει γίνει αυτό το πέρασμα και στον τομέα των μεταφορών, όπου μιλάμε για επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα ή με σοβαρές αναπηρίες. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πού και πώς κινούμαστε, αλλά ως προς το θέμα αρχής συμφωνούμε και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν αυτά τα μέτρα που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Γεζίνα Μάισνερ. Ναι. ευχαριστώ. Εκπροσωπώ εδώ πέρα την Ιζασκούν Μπιλμπάου γενικά θεωρώ πως είναι θετικό το ότι ασχολούμαστε με αυτό το θέμα γιατί μεγαλώνει το ποσοστό ατόμων με αναπηρία γενικώ στον πληθυσμό και βεβαίω η προσβασιμότητα βοηθάει, ξέρω εγώ, και μία μητέρα με καροτσάκι. Λοιπόν, θα διαβάσω τα αγγλικά. Καλωσορίζουμε αυτή την πρωτοβουλία για να φύγουν όλα τα εμπόδια για τους πολίτες μας στην εσωτερική αγορά. Αυτό πρέπει να γίνει σε στενή συνεργασία με τις ενώσεις επιβατών, τους χρήστες και τον κλάδο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πρόσβαση στις υποδομές σε επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα ή άτομα με αναπηρία. Πέρα από την ανάγκη να βελτιωθεί η πρόσβαση στους διάφορους τρόπους μεταφοράς και στις υποδομές θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να διασφαλιστεί μια καλύτερη προσβασιμότητα στα site ε, και στα συστήματα πληροφορική. Ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, μεγάλο ποσοστό των υπηρεσιών πολλούνται μέσω διαδικτύου. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένα εργαλεία για να διευκολύνουμε την ε, προσβασιμότητα των μέσων μεταφοράς. Και αναμένω βεβαίως να ε, συνεργαστώ με τους ηγητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρή Κριστίν Νότριου. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την Επιτροπή, καθώς και τον εισηγητή. Θα ήθελα να είμαστε πραγματιστές σε θέματα αναπηριών, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο όλοι προσπαθήσατε να βρεθείτε σε σταθμούς με ένα παιδί με αναπηρία, που βρίσκεται σε αναπηρική ε, καρέκλα και πρέπει να κυκλοφορήσει έτσι. Εγώ για 33 χρόνια που ζω στη Γαλλία μπορώ να σας πω ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Αυτή η πρόταση οδηγίας θα πρέπει να ε, επιταχύνει αυτή την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. Θα πρέπει όμως πραγματικά να βελτιωθεί μέχρι τώρα. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν φτάσαμε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Νομίζω, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει σαφήνεια, και το είπατε κι εσείς, σε σχέση με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα στο πεδίο εφαρμογής, δεν αποτελούν ένα ε, σωστό βήμα μέσα στα πλαίσια μιας ενωμένης Ευρώπης και στα πλαίσια της δημοκρατικής νομιμότητας. Επίσης μιλάμε για εισαγωγή συνάφειας και συνέπειας μεταξύ των κανόνων που ισχύουν στις ΕΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό με ανησυχεί γιατί δεν βλέπετε ή κάνετε ότι δεν βλέπετε ότι πέρα από το συμβολικό χαρακτήρα ε, του να συμβαδίζουμε με την νομοθεσία των ε, ΗΠΑ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις αμερικανικές επιχειρήσεις οι οποίες ε, ακολουθούν αυτούς τους κανόνες, άρα δεν θα έχουν ένα επιπρόσθετο φόρτο όπως θα έχουμε εμείς, δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Μιλήσατε για τις εξαιρέσεις για τις ε, μικροεπιχειρήσεις αλλά αυτό ε, δεν μπορεί να αντισταθμίσει την κατάσταση ιδιαίτερα στη Γαλλία. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η ΤΙΖΑ και το TTIP δεν βρίσκουν σύμφωνο τους Ευρωπαίους πολίτες επί του παρόντος. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή τη συλλογιστική που διέπει την οδηγία. Και επίσης μιλάμε για τα ΜΕΑ, βεβαίως θα πρέπει να ορίσουμε εκ νέου τις αναπηρίες, για τις εγγύους άλλα είναι τα προβλήματα, άλλα θέματα προσβασιμότητας, αλλά δεν πρέπει να τα βάλουμε όλα στο ίδιο σακί, γιατί τότε δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Ευχαριστώ για την Κομισιόν και πάλι η κυρία Πλασανσία. Ωραία. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να απαντήσω στα βασικά στοιχεία τους. Όπως τα σημείωσα εγώ. Κάποιες από τις ε, παρεμβάσεις είπαν ε, πώς ε, σχετίζεται αυτή η οδηγία με την, την υπόλοιπη υφιστάμενη νομοθεσία για τις μεταφορές. Να ξεκαθαρίσω πως οι σχέση τους είναι συμπληρωματικοί. Τα στοιχεία που καλύπτει η διάταξη περί προσβασιμότητας ε, στο διαδίκτυο, τα εξμεστήρια, τηλεφορία σε πραγματικό χρόνο, μηχανήματα έκτοσης εισιτηρίων και μηχανήματα αυτοεξυπηρέτησης δεν αναφέρονται σε μεγάλο βαθμό στο υπόλοιπο υφιστάμενο ευρωπαϊκό δίκαιο. Η οδηγία επίσης αναφέρεται στην εναρμόνιση της, στην δυνατότητα των κρατών μελών να αποφασίσουν να εναρμονίσουν. Είναι μια επιλογή, είπαμε. Αυτό σημαίνει πως στην μόνη περίπτωση στην οποία υπάρχουν απαιτήσει περί προσβασιμότητας μεταφορές, δηλαδή στους σιδηροδρόμους, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Η οδηγία δεν καλύπτει άλλους τομείς όπως τα οχήματα, παραδείγματος χάρη, δεν επιβάλλει άμεσες Υποχρεώσει στους κατασκευαστών οχημάτων γιατί υπάρχει ήδη, υπάρχουν ήδη άλλε διατάξει. Οπότε η οδηγία αυτή συμπληρώνει υφιστάμενο ευρωπαϊκό δίκαιο. Όταν ε, λέμε το ποιο θα ωφεληθεί από αυτό, βεβαίω, η οδηγία χρησιμοποιεί τον όρο άτομα με περιορισμούς ε, στη λειτουργικότητα και άτομα με αναπηρία. Ο ορισμός των ατόμων με αναπηρία είναι αυτός της σύμβασης του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία και το σκεπτικό πίσω από την έκφραση λειτουργική περιορισμή είναι για να καλύψουμε άτομα με προσωρινούς περιορισμούς γιατί η σύμβαση περί αναπηρίας απαιτεί να είναι μακροχρόνια ε, η αναπηρία ή ο περιορισμός αλλά κάποια αυτά άτομα. Είχε κάποιος που έχει σπάσει το πόδι του. Ε, ή προσωρινά δεν μπορεί να δει μετά από μια εγχείρηση. Όλα αυτά τα άτομα δεν είναι άτομα με αναπηρία, αλλά θα ωφεληθούν από την προσβασιμότητα που θα θέσει ενισχύει η οδηγία. Επίσης, ο νόμος περί προσβασιμότητας συμπληρώνει τους σχετικούς κανονισμούς για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα στις μεταφορές με στόχο την ε, βοήθεια. Στόχος εδώ πέρα είναι να υπάρχει ίση πρόσβαση. Για να υπάρχει ίση πρόσβαση χρειάζεται, χρειάζονται και τα δύο. Και προσβασιμότητα και βοήθεια. Αυτά πάνε μαζί και όσο περισσότερη προσβασιμότητα υπάρχει, τόσο περισσότερο θα μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί ανεξάρτητα τις υπηρεσίες και με λιγότερη ανάγκη βοήθειας. Αλλά βέβαια η βοήθεια παραμένει. Και δεν υπάρχει ανάγκη να μεταρρυθμίσουμε την υπόλοιπη νομοθεσία. Οπότε, επιβεβαιώνω πως ε, πράγματι ε, πλήρει αυτό τις απαιτήσει ε, περί βοήθειας. Λοιπόν, ε, σίγουρα προσπαθώ να δω ποια ήταν η επόμενη ερώτηση. Σε σχέση με τη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους. Είχαμε εκτεταμένες ε, διαβουλεύσεις επίσης και συζητήσεις με διάφορους ενδιαφερομένους, άτομα με αναπηρίες κτλ. Υπάρχει επίσης ε, μια σχέση μεταξύ αναπηρίας ε, και γύρατος. Ε, δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην εμπίπτουν οπωσδήποτε στον κλασικό της αναπηρίας, αλλά μπορεί να υπάρχει βαρικοία, μια δυσκολία στην κίνηση κτλ. και την όραση, οπότε υπάρχει αυτή η σχέση και θα συνεχίσουμε να έχουμε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους. Όταν μιλάμε λοιπόν Τώρα για το θέμα την, της ευθυγράμμισης με τις ΙΠΑ. Να ξεκαθαρίσω. Εδώ πέρα βασιζόμαστε στο μοντέλο νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς. Είναι ένας ευρωπαϊκός τρόπος ε, ρύθμισης. Διορίζουμε δηλαδή, κάποιες γενικές αρχές ε, λειτουργικών απαιτήσεων και μετά έχουμε κάποιες ευρωπαϊκές διατάξεις που με έναν τρόπο εθελοντικό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια συμμόρφωση. Η ευθυγράμμιση λοιπόν που αναφέρεται στο μνημόνιο το σχετικό είναι για να έχουμε κάποιες ε, παγκόσμιες προδιαγραφές ε, σε σχέση με την τεχνολογία της πληροφορικής ε, και των τηλεπικοινωνιών. Το είδαμε αυτό και στην οδηγία για την προσβασιμότητα στις ιστοσελίδες του δημοσίου τομέα, όπου υπήρχε μια έκκληση να χρησιμοποιηθούν οι παγκόσμιες, ε, κάποιες παγκόσμιες απαιτήσει προσβασιμότητας. Όταν μιλάμε λοιπόν για εναρμόνιση σε παγκόσμιο επίπεδο, μιλάμε για τις ιστοσελίδες. Θα ήθελα λοιπόν να τελειώσω με αυτά. Νομίζω ότι κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις. Αλλιώ είμαι βεβαίως στην διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ντάβος Κέλετς και πάλι Ντάβορ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις για τα πολύ χρήσιμα σχόλια και τα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ και την εκπρόσωπο της Κομισιόν γιατί μας έδωσε λεπτομερείς ε, απαντήσεις. Ξέχασα να αναφέρω ότι η ΙΜΚΟ είναι η υπεύθυνη επί της επιτροπή και εμείς θα εκφράσουμε την άποψή μας στα τμήματα της οδηγίας που ε, είναι βρίσκονται υπό δική μας αρμοδιότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες και τους κοιόδης. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank. Und der Ευχαριστώ. Το σχέδιο της νομοδοτήσεως θα υποβληθεί τον Νοέμβριο. Λέει ο Πρόεδρος Κράμερ. Και τώρα θα προχωρήσουμε στο θέμα υπαριθμών 7 της ημερησίας διατάξεως στρατηγική αερομεταφορών στην Ευρώπη. Εδώ έχουμε ο τον κύριο Παύλ Τέλιτσκα. Εδώ και δέκα μήνες ε, ξέρετε ότι όπου από την Επιτροπή, από πλευράς ε, Επιτροπής έγινε η παρουσίαση της στρατηγικής για τις ε, αερομεταφορές από τον ε, Επίτροπο Μπούλς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς αντιλαμβανόμαστε το θέμα και από πλευρά σκιωδών και θα ήθελα να πω ότι βρίσκομαι πάντα σε στενή επαφή με τους συναδέλφους, εξέφρασα τη δική μου συλλογιστική και οι συνάδελφοι έκαναν σχόλια τα οποία έλαβα υπόψη. Όπως είπαμε και με τους σκιώδεις, δεν θέλουμε να επαναλαμβάνουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής. Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τα σημεία κλειδιά και να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν στο προσχέδιο της Επιτροπής. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλά σημεία κλειδιά στην έκθεση αυτή και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη καταρχήν ότι οι αερομεταφορές είναι ένας τομέας όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις και αυτό που έχει σημασία είναι πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε ποια είναι η εμπειρία μας και ποιο είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα της προσέγγισής μας. Θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το πρότυπο των ευρωπαϊκών αερομεταφορών και αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν θα πρέπει να δεχτούμε τις πιέσεις που προϋπάρχουν, αλλά να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια με βάση τις ανάγκες της αγοράς και τις παροχές της αγοράς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που θα ήθελα να τομίσω, το, να τονίσουμε, συγχωρείτε. Επίσης, ε, θα ήθελα να δούμε τους σχετικούς δείκτες, γιατί αυτό που έχει μεγάλη σημασία για τον τομέα είναι όχι να δούμε τι θα είναι οι αερομεταφορές το 2030, αλλά να έχουμε μία μακροχρόνια ε, θεώρηση για να γίνει προγραμματισμός και οι σχετικές επενδύσεις. Νομίζω ότι αυτός ο, ο δείκτης συνδεσιμότητας είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης για να δούμε ποια είναι η δυναμική και οι δυνατότητες του τομέα. Η συνδεσιμότητα δεν αφορά την συχνότητα, την ένταση, τον χρονισμό, αλλά θα πρέπει να σχετίζεται και με τις ευκαιρίες που έχουμε σε σχέση με το περιβάλλον, με τις περιπτώσεις πολύ υψηλής κυκλοφορίας, στενοπών κλπ. Όπως ξέρετε, είμαστε και η μεγαλύτερη αγορά και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί γιατί θα υπάρχει και καλύτερη συνδεσιμότητα και μεγαλύτερες ευκαιρίες. Το θέμα της ασφάλειας επίσης είναι ύψης της σημασίας. Ξέρετε τι αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια. Νομίζω ότι οι προκλήσεις θα είναι και πολύ μεγαλύτερες, καθώς και κίνδυνοι. Θα πρέπει να βασιστούμε στις πληροφορίες και στις νέες τεχνολογίες, καθώς και σε μοντέλα, σε πρότυπα ε, παγκόσμιας εμβέλειας θα πρέπει να δούμε και θέματα ελέγχου, και οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν και ακόμα μεγαλύτερες ε, ε, ευκολίες, ξεκινώντας από το pre-check-in και ούτω καθεξής. Μιλάμε για την ε, ευρωπαϊκή λεωφόρο των εθέρων. Το βλέπουμε στον κανονισμό του 2004, τον κανονισμό 551, όπου υπάρχουν και οι τεχνικές προδιαγραφές και νομίζω ότι η, η διευρωπαϊκή λεωφόρος των εθέρων θα πρέπει να ισχύει στους εθέρες όπως ίσχυε και στις ε, οδικές μεταφορές. Τέλος, ε, είμαι σίγουρος ότι θα έχετε πολλές ερωτήσεις και ίσως θα θέλετε να δούμε ζητήματα σε περισσότερη λεπτομέρεια. Θα υποβάλω και εγώ τροπολογίες, δικές μου τροπολογίες. Θα ήθελα να μιλήσουμε και για συμφωνίες αερομεταφορών ή αερομεταφορών γενικότερα Πιστεύω ότι θα βρείτε στην ε, έκθεση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τον τομέα και νομίζω ότι θα έχουμε και μία νέα ε, εμπειρία με βάση τα συμπεράσματα στα οποία θα φτάσουμε. Θα μπορούσα να μιλήσω περισσότερο και να μιλήσω για το TNT, για τις πολυτροπικές μεταφορές, για τα κομβικά αεροδρόμια, αλλά αυτό θα ήθελα να μας απασχολήσει και στο μέλλον σαν ολοκληρωμένος τρόπος μεταφοράς. προβάλλοντας και τα περιφερειακά αεροδρόμια δηλαδή να, δούμε, να τα δούμε όλα με στα πλαίσια του ten Πιστεύω ότι επειδή λάβατε έγκαιρα την έκθεση, την έχετε μελετήσει σχετικά και περιμένω τις παρατηρήσεις σας έτσι ώστε το έγγραφο αυτό να γίνει πιο ολοκληρωμένο και να υποβάλουμε προτάσεις αργότερα και προς την Κομισιόν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεση, λέει η κυρία Κλούν. Και χαίρομαι γιατί με συμπεριέλαβε και εμένα στα σχόλιά του. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία με βρίσκουν σύμφωνοι. Θεωρώ ότι οι αερομεταφορές θα πρέπει να ολοκληρωθούν καλύτερα τα επόμενα 20-30 χρόνια γιατί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικονομίας και φυσικά υπάρχει και το θέμα του κόστους των ε, περιορισμών και του γεγονότος ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί με βάση και εξωγενείς παράγοντες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την αυξητική πορεία των αερομεταφορών. Μιλάμε για μια αύξηση 5% τα επόμενα χρόνια και μιλάμε για μια, ε, ένα συνολικό μερίδιο δικό μας της τάξης του 40%. Θα πρέπει λοιπόν και τα Εθνικά Κοινοβούλια να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε ε, ενδεχόμενους ανταγωνιστές, αλλά να τους αντιμετωπίσουμε. Ως προς τις ε, διευρωπαϊκές, τη διευρωπαϊκή αυτή λεωφόρο στις αερομεταφορές είναι πολύ ε, σημαντική γιατί οι απεργίες στήχησαν τα τελευταία χρόνια 9,5 δις ευρώ, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και αυτή την πτυχή του θέματος θα πρέπει να προχωρήσει και ο Ευρωπαϊκός Ενιαίος Ουρανός. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάπως να αντιμετωπίσει και αυτό το θέμα. Ως προς το δίκτυο συνδεσιμότητας είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για τον εισηγητική και για όλους μας, διότι θα πρέπει να είναι ε, μετρήσιμη αυτή η συνδεσιμότητα. Έγιναν πολλές συζητήσεις σε αυτή την ε, Επιτροπή. Θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τα περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία θα πρέπει να έχουν μία μορφή συνθεσιμότητας. Και το θέμα της ασφάλειας ε, είναι στο προσκήνιο. Θα πρέπει να είμαστε πιο ευφυείς σε θέματα ασφάλειας, να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα ορίζεται και ο έλεγχος διαβατηρίων. Θεωρώ ότι τα διαβατήρια θα πρέπει με βάση τα βιομετρικά δεδομένα να είναι πιο σίγουρα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται ε, επιπρόσθετη ασφάλεια υποτύπου υποδομών. Έχει μεγάλη σημασία επίσης να δούμε και το θέμα του περιβάλλοντος και και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα να προσθέσω και μερικά στοιχεία, αλλά δέχομαι με την όθηση που δίνει στο θέμα των αερομεταφορών και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή η οποία ολοκληρώνει το πακέτο το οποίο ζητούσαμε ασμένος εδώ και πολύ καιρό. Και ε, εδώ μιλάμε για έναν τομέα ύψης της σημασίας στα πλαίσια της παγκόσμιας κακέρας και για την ε, παγκόσμια ε, οικονομία. Και αυτό αφορά και τις ε, θαλάσσιες μεταφορές, οδικές, αλλά ιδιαίτερα τις αερομεταφορές. Θα ήθελα να τονίσω ότι η γενική πρόταση συνδέει διάφορα επιμέρους ζητήματα. Εμείς θεωρήσαμε ότι τη στιγμή που έχουμε τα τομεακέ, τομεακά πακέτα, τα πολυτροπικά, θα θέλαμε να υπάρχει ευελιξία και εξυγχρονισμός και στον τομέα των αερομεταφορών. Κάτι το οποίο δεν είχαμε κάνει σε λεπτομερία. Θα πρέπει να τον εντάξουμε στο κοινωνικό πακέτο να τονίσουμε την ε, υποστήριξη της ε, Κομισιόν μέσω μιας ε, πλατφόρμας για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, την αναγνώριση της εργασίας των εργαζομένων, τη διαδικασία πιστοποίησης και αδειοδότησης, τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και την ε, προσωρινή εργασία και την επισφαλή εργασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρχαν, υπήρξαν πολλές επιπτώσεις με την επισφαλή εργασία, κάτι το οποίο είχε επιπτώσεις και στο κοινωνικό πακέτο. Να δούμε πώς οι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν το θέμα της απασχόλησης. Ως προς τους επιβάτες, τα δικαιώματα των επιβατών, θα δούμε τι θα εγκρίνει το Κοινοβούλιο με βάση την ανάγνωση που έχει γίνει και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εθνικοί αερομεταφορείς οδήγησαν και στη, σε πολλές επιχειρήσεις ε, εταιρείες χαμηλού κόστους. Και γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύονται τα δικαιώματα των επιβατών, γιατί πολλές φορές αμφισβητήθηκαν τα ε, δικαιώματά τους λόγω χαμηλού κόστους και εταιριών low cost. Γι' αυτό θα πρέπει να υπερασπιστούμε τους επιβάτες και τα δικαιώματά τους, γιατί από αυτό εξαρτώνται και άλλες δυνατότητες. Βλέπουμε πολλές αλλαγές και προβλέψεις σε σχέση με τις νέες προσφορές των εταιριών low cost θα πρέπει να δούμε και τον ψηφιακό τομέα, τις ψηφιακές εξελίξεις. Θα πρέπει οι νέες τεχνολογίες να είναι φιλικές προς τον χρήστη με βάση τις δυνατότητες, τις διευκολύνσεις και τις ευελιξίες, τη γενικότερη ευελιξία και προσβασιμότητα και ως προς τις υποδομές θα πρέπει και πάλι να κινηθούμε προς αυτές τις ε, δυνατότητες γιατί πολλές φορές ε, στα πλαίσια της αντιμετώπισης, αντιμετώπισης της κρίσης ε, δημιουργήθηκαν άλλα δεδομένα και δυστυχώς δεν ήταν, δυσ... δεν ήταν εύκολο να τα εντάξουμε όλα αυτά και να τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, κομβικά αεροδρόμια, τα οποία αντιμετωπίσαμε διαφορετικά από τα περιφερειακά. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν, τι ορίζοντες ανοίγουν. Δεν θέλουμε μακροαεροδρόμια όπου τεράστια αεροδρόμια όπου θα πρέπει να διανύσει χιλιόμετρα ο επιβάτης μέσα σε αυτά τα τεράστια μολ αλλά θα πρέπει να ε, υπάρχουν κλάστερ περιφερειακών αεροδρομίων τα οποία και θα πρέπει να προωθήσουμε ανάλογα. Και αυτό αφορά και τον τομέα του κάρκου. καθώς και τις υπερπτήσεις που γίνονται κατά τις νυχτερινές ώρες. Θα πρέπει να δούμε ποιες δυνατότητες διανοίγονται υπομορφή κλάστερ και μέσα στα πλαίσια φυσικά και των ε, εκπομπών. θα πρέπει να δούμε και την τιμολόγηση των υπηρεσιών, αλλά να δούμε πώς θα συνδέσουμε και τις αερομεταφορές με τη μείωση των εκπομπών. Τζάκι Φώστερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό πάρα πολύ καλά, συντονιστήκαμε, συναντηθήκαμε και βεβαίως ε, έχει και μία ιδέα μετά ε, για το τι θέλουν οι σκιώδεις εισηγητές. Και καλό είναι αυτό νομίζω. Και πραγματικά το έγγραφο ε, που συνέταξε ο κύριος Τελίτσκα σε γενικές γραμμές αντικατοπτρίζει πολλές απόψεις ε, των σκιωδών και λοιπόν. Νομίζω λοιπόν πως ε, είναι κατάλληλη η στιγμή, γιατί είμαστε τυχεροί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη θα έλεγα. Έχουμε πολύ ανταγωνιστικό κλάδο, δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας. Διαφωνώ με την κυρία Γιάλα Σέντερο σε έναν βαθμό, είναι η πιο ρυθμιζόμενη ε, μορφή μεταφορών και ισχύουν οι κανονισμοί για όσους εργάζονται σε αυτόν τον κλάδο σε κρίσιμες θέσεις. Δεν υπάρχουν έτσι κάποια ε, συμβόλαια που δεν ρυθμίζονται. Ρυθμίζονται πάρα πολύ και έτσι θα πρέπει να είναι άλλωστε. Υπάρχουν βεβαίως διαφορές γιατί υπάρχει και εποχιακή εργασία στον τομέα των τσάρτερ αλλά σε γενικέ γραμμέ νομίζω πω οι δουλειέ ε, και το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό και γι' αυτό δεν φεύγει κανεί από τον κλάδο και αυτό είναι καλό σημάδι. Η οικονομία ωφελείται και νομίζω αυτό το οποίο είπε ο κ. Σταλίτσκα ε, για την εφοδιαστική αλυσίδα είναι ότι εμείς είμαστε σε παγκόσμια ηγετική θέση στην κατασκευή αεροσκαφών και τα αγοράζουν και οι δικές μας αεροπορικές εταιρείες και συχνά αυτό δεν το παρατηρούν τα μίμια και όσοι ασκούν κριτική. Και βεβαίως αυτό μετά έχει σχέση και με το περιβάλλον, γιατί ε, και εδώ πέρα παίζουμε ηγετικό ρόλο, είχαμε τους καθαρούς ουρανούς 1, 2 και πάλι βλέπουμε ακριβώ ε, το πώς αντιμετωπίζουμε τα περιβαλλοντικά ζητήματα της αεροπορίας και είμαστε χρόνια μπροστά από άλλους. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και βεβαίως αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από το Μοντρεάλ. Οπωσδήποτε στηρίζουμε ένα παγκόσμιο σύστημα, αλλά όχι παράλληλα με την παλιά ιδέα, γιατί έτσι δεν θα λειτουργήσει. Τώρα περιμένουμε τον Οκτώβριο. Για αυτά τα οποία είπατε επίση για τον ανταγωνισμό. Μ' αρέσει η προσέγγιση του εισηγητή γιατί ανταγωνισμός δεν σημαίνει προστατευτισμός. Η πρόσβαση στην αγορά έχει ωφελήσει πολύ τον καταναλωτή μαζί με την απελευθέρωση και αυτό το οποίο είπαμε για την ασφάλεια και κυρίως το πόσο εξελιγμένες θα είναι οι πρακτικές ασφαλείας. Ε, έχει μεγάλη σημασία γιατί το κόστος ε, για τον καταναλωτή και τον κλάδο ε, γίνεται όλο και πιο μεγάλο. Και οι ιδέες αυτές που έχουν δοκιμαστεί στη ΣΥΠΑ και αλλού νομίζω αξίζει να τις εξετάσουμε είτε μιλάμε για προεγγραφή είτε για οτιδήποτε άλλο. Τώρα για το πού μπορούμε να πάμε από εδώ και μπρος. Νομίζω σωστά αναφέρουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Το θέμα στο ευρωπαϊκό το ότι έχουμε κολλήσει εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο είναι δικαιολογία. Τα κράτη-μέλη το χρησιμοποιούν ως δικαιολογία. Και εμείς προχωρούμε με το ΣΕΖΑΡ και μπορούμε και με την αναδιάρθρωση του εναερίου χώρου. Δεν υπάρχει λόγος να κολλήσουμε και πρέπει να προχωρήσουμε γιατί αλλιώ θα υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο για όλου. Αλλά το θέμα είναι τελικά εάν θέλουμε να προχωρήσει αυτό ο κλάδο όσο χρειαζόμαστε να προχωρήσει και βεβαίω να δημιουργήσουμε ε, και την απαιτούμενη δυνατότητα. Υπάρχουν πολλέ αντιρρήσει στα κράτη-μέλη και πάρα πολλά έργα σταματάνε γιατί ο κόσμο δεν θέλει παράδειγμα του χάρη να έχουν ένα διάδρομο όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και εάν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτό τότε ο κλάδος στην Ευρώπη θα μειωθεί και τότε θα πάνε σε τρίτες χώρες οι επιχειρήσεις. Αν αυτό θέλετε, καλώς. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θέλω εγώ και δεν νομίζω πως είναι αυτό που θέλει και η Επιτροπή. Εάν θέλουμε λοιπόν ανάπτυξη, πρέπει και τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν το νου και την πολιτική βόληση να λάβουν τις αποφάσεις που θα φροντίσουν να είμαστε επιτυχείς στο μέλλον. Συνολικά λοιπόν νομίζω πως είναι εξαιρετική η έκθεση. Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα, λίγα πράγματα για αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής και αυτά τα οποία βλέπουμε μέχρι στιγμής και προφανώς ε, εξετάσαμε τις δύο γνωμοδοτήσεις. Κάποια κομμάτια του τάξη είναι καλά, αλλά σε γενικές γραμμές είναι νομίζω μια εξαιρετική έκθεση κύριε εισηγητά και σας ευχαριστώ που την ε, δεχτήκατε και που κάνατε τόσο καλή ε, δουλειά. Και οπωσδήποτε εμείς στο ECR σας στηρίζουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ντάβος Κέρλιτς. Ντάβος Κέρλιτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, βλέποντας την εξέλιξη της αεροπορίας σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως είπε η κυρία Φώστερ, πρέπει να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αεροπορίας. Όμως πρέπει να γίνει με τρόπο βιώσιμο και να λάβουμε υπόψη την ε, κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποσχεθεί εδώ πέρα να παίξει έναν ηγετικό ρόλο. Η κυρία Ταλίτσκα έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης, ο κύριος Ταλίτσκα, και τον ευχαριστώ γιατί έχει λάβει υπόψη όλα τα σημαντικά στοιχεία. Συμφωνώ με το θέμα της συνδεσιμότητας, γιατί ο εισηγητής τονίζει το ζήτημα της διαλειτουργικότητας ως το μόνον τρόπο για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της αεροπορίας. Επίσης, η διαλειτουργικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και αυτό φαίνεται στην έκθεση. Η έκθεση Επίσης αναφέρει ότι θα πρέπει να δούμε το δίκτυο των ε, δύο Ευρωπαϊκών δικτύων. Θα πρέπει να υπάρξει αυτό ακριβώς για να μπορούν να μετακινηθούν οι επιβάτες από το ένα μέσο στο άλλο και θα πρέπει να προωθήσουμε την χρήση των σιδηροδρόμων ως εναλλακτική στα αεροπλάνα. Όσον αφορά τώρα την επιβατική κίνηση, θα πρέπει να επιμείνουμε στα δικαιώματα των επιβατών, των αεροπορικών επιβατών, ειδικά όταν μιλάμε για πρόσβαση ε, για όλους τους Ευρωπαίους και να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για να είναι προσβάσιμη η αεροπορία στα άτομα με αναπηρία. Τώρα, Βλέπουμε τώρα πως ο κλάδος είναι απορριθμισμένος και έχει βεβαίως την πίεση που υφίσταται, πολύ χαμηλές τιμές. Πρέπει να δούμε και το καθεστώς των εργαζομένων και πώς μπορεί κάτι τέτοιο να επηρεάσει την ασφάλεια των πτήσεων την ποιότητα των υπηρεσιών και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ένα από τα στοιχεία που τράβηξε την προσοχή μου είναι η κυκλική οικονομία. Εκεί όπου λέει δηλαδή ότι το πακέτο της ε, Κομισιόν ε, για την κυκλική οικονομία θα πρέπει να το δούμε υπό το πρίσμα της μείωσης των ε, εκπομπών στα αεροπορία ειδικά κατά την άφηξη ε, και την ε, αναχώρηση από αεροδρόμια. Θα ήθελα λοιπόν ο κύριος Τέλητσκα εδώ να το ξεκαθαρίσει αυτό το κομμάτι της έκθεσης. Όσον αφορά τώρα την βιωσιμότητα, η Ευρώπη πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο και να αποτελέσει παράδειγμα βιώσιμης ε, αεροπορίας. Ε, πρέπει να μειώσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο της αεροπορίας και να ενισχύσουμε τη μάχη κατά της ε, κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι μόνο θέμα διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και άλλων αερίων του θερμοκηπίου και αυτών με τα σωματίδια που αποτελούν κίνδυνο για την υγεία. Οπότε το ζήτημα της ποιότητας του αέρα αφορά ε, τη δημόσια υγεία. Οπότε πρέπει η αεροπορία να βασίζεται στην αεφορία, να επενδύσουμε στην έρευνα και την καινοτομία και υποστηρίζω τη συμπερίληψη εναλλακτικών καυσίμων και βεβαίως υπάρχει και το θέμα των λοιπόν τεχνολογιών, η ανάπτυξη νέων κινητήρων που θα εκπέμπουν λιγότερο ε, επίσης, πρέπει να έχουμε κατά νου αυτούς ε, που ζουν σε υψηλότερα μέρη, υποφέρουν από τον θόρυβο των αεροπλάνων. Μιλάμε για πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που ζουν κοντά σε αεροδρόμια. Αυτά ήθελα να αναφέρω και ελπίζω στο μέλλον να ξεκαθαρίσουν αυτά τα ζητήματα μέσω της συνεργασίας και με τον κύριο Τέλιτσκα. Ευχαριστώ η Μαρή Κριστίνα Νοτέ. Ευχαριστώ ε, και εσάς κύριε Σιγητά. Ακούγοντάς σας κύριε Τελίτσκα λέτε δηλαδή ότι ο τομέας των ε, της αεροπορικής μηχανής είναι πιο επιτυχημένος. Ναι, είναι όμως και επιτυχία άραγε του ελεύθερου ανταγωνισμού που τόσο λατρεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κοιτάζω τα τελευταία 30 χρόνια. Η κατάσταση είναι διαφορετική. Από την απελευθέρωσή της που άρχισε η δεκαετία του 80 πάντοτε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υφίσταται τις συνέπειες των όσων τεκταίνονται είτε στον Πακού είτε στον Πρισσικό κόλπο οι ευρωπαϊκοί φορείς έχουν στην ουσία ε, απομακρυνθεί από τις γραμμές που συνδέουν την Ευρώπη με την ε, Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει την αγορά της στον ανταγωνισμό, δεν μπόρεσε όμως να τοποθετήσει τις εθνικές της εταιρείες στις ε, αγορές αυτές που ανοίγουν και αυτές και οι ευρωπαϊκές εταιρείες δηλαδή μόλις και που επιβιώνουν. Το ίδιο και η France KLM. Πρόσφατα, σε έκθεσή της η Γαλλική Γερουσία είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει να πετούν όλο και περισσότερα αεροπλάνα αλλά σε ξένο ουρανό τελικά. Αυτά λέει η Γερουσία. Αυτά που επιβάλλει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, μη επιβάλλοντας μη επιβάλλοντα στου επενδυτέ και τις επενδύσει από τρίτε χώρε δεν επιτρέπονται. Για παράδειγμα, η Αλιτάλια, αρκετά εύκολο παράδειγμα, η εταιρεία Etihad έλαβε την άδεια να πράξει αυτά που δεν επέτρεψαν στην Ιταλική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις ε, ρυθμίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις λόγω αυτών των ρυθμίσεων. γιατί η Ρωσία τώρα η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι καμιά επιτυχία, οδηγεί στην αβεβαιότητα την απασχόληση και μειώνει την ανταγωνιστικότητα. Το ίδιο όπως και η ψευδοανεξάρτητη, το pay to fly, οι ε, συμβάσεις με μηδενικό χρόνο και ούτε Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών, λίγο ότι οι ξένες εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να αποζημιώνουν, για παράδειγμα, του επιβάτε σε περίπτωση καθυστερήσεων. Τα μέτρα που προβλέπει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου φαίνονται μη ικανοποιητικά για την εξασφάλιση του πλήρου ανταγωνισμού στον τομέα των ενεργειών μεταφορών, διότι αυτό υποτίθεται ότι είναι ο στόχος μας, στρατηγικό. Στην έκθεση λένε ότι ο προστατευτισμός δεν αποτελεί ποτέ λύση και οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανοιχτή αγορά για να μπορέσουν να ανθίσουν. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλο σφάλμα. Και παραδόξως οι, Ευρω... δεν έχουν ανοίξει την αγορά τους. Και αυτός ο... αυτά τα λόγια, πολύ φιλελεύθερα υποτίθεται, ωστόσο οι Αμερικανοί ενισχύουν τις εξαγωγές τους και προστατεύουν τους στρατηγικούς τους τομείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, έχει θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο λειτουργεί αντίθετα με τα συμφέροντα των εταιριών, τους, των εταιριών της. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθεί προς μια προστατευτική κατεύθυνση και ιδίως η 868 του 2004 για τον αφέμητο ανταγωνισμό και 1008 του 2008 για τον έλεγχο των ευρωπαϊκών εταιριών. Το ίδιο στις συνομιλίες με τρίτες χώρες για τις οποίες έχει λάβει ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντολή και όπου θα ήθελα πολύ οι χώρες μέλη να μπορούν να ελέγχουν τι κάνει, θα πρέπει αυτή η προσέγγιση να επιβληθεί οπωσδήποτε. Εν συμπεράσματι, οι στόχοι που περιλαμβάνει το έγγραφο της Κομισιόν και το οποίο εσείς χαιρετίζετε κύριε ε, εισηγητά, μου φαίνονται απλό ευχολόγιο. Θα υποβάλουμε βεβαίω τροπολογίε για να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε μαζί και να προχωρήσουμε προς μια συγκεκριμένη στρατηγική και όχι μια στρατηγική η οποία απλώς διακατέχεται από καλές προθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Επτά μου μένουν εγγεγραμμένοι, αλλά ο χρόνος ε, μας τελειώνει, γι' αυτό θα ε, κλείσω τώρα και θα σας δώσω για 1,5 λεπτό τον λόγο ο κ. Κόχ. Ευχαριστώ κύριε Τέλιτσκα πρώτα για την εξαιρετική σας έκθεση που σωστά ε, σημειώνει τα κέντρα βάρους της προτάσεως της Κομισιόν, ίσως ορισμένα κάπως ε, να χρειάζονται περισσότερη επεξεργασία της αυτό έχει σχέση και με τους περιορισμούς που ισχύουν για το κείμενό σας. Βεβαίω, ε, εσεί μιλήσατε ήδη για τις συμφωνίες για τι ενεργέ μεταφορέ. Ω εισηγητή του Λαϊκού Κόμματος για την ε, γνωμοδότηση στην ΕΜΠΛ, θα συνεργαστώ μεταξύ σα, θα κάνω προτάσεις. Έχουμε 118 τροπολογίες. Θα γίνει την επόμενη εβδομάδα η πρώτη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και ε, αναμένω τη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να αναφέρω στη συνάδελφο ότι μάλλον μπερδεύεται την περίπτωση της Αλιτάλια με την Έφιαντ, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν αναγνωρίστηκε η, δεν αναγνωρίστηκαν οι κρατικές ενισχύσεις, άρα όλα έγιναν καλώς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τέλισκα γιατί το θέμα είναι άκρος ενδιαφέρον και συμμερίζομαι την προσέγγιση του, αλλά το βασικό είναι ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός. Υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να πω ότι ίσως υπάρχουν και διμερεί ζητήματα μεταξύ κρατών, όμως το ζήτημα αυτό δεν επιλύεται γιατί υπάρχει και το θέμα του Γιβραλτάρ. Είναι ευρωπαϊκός χώρος και γι' αυτό θα πρέπει να επιλύσουμε το ζήτημα. Διαφορετικά δεν θα υπάρχουν ε, θετικές επιπτώσεις ως προς το περιβάλλον, τους ναύλους και ούτω καθεξής. Ε, μιλάμε για 800 εκατομμύρια περίπου επιβάτες που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Ένα άλλο ζήτημα είναι οι κρατικές ενισχύσεις, το οποίο βλέπουμε στο σημείο 12 της έκθεσης. Θα είμαι σύντομη. Μιλάμε για εδαφική συνοχή και κρατικές ενισχύσεις. Η καλύτερη λύση θα ήταν να φτάσουμε στο πρώτο ε, σκέλος της δημόσιας διαβούλευσης έτσι ώστε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουν και το θέμα των εμπορικών συμφωνίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ματίας Φων Μίλτεμπεκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ βέβαια, να ευχαριστήσω τον κύριο Τέλετσκα, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα που πρέπει να ακουστούν σε αυτή την έκθεση. Πρώτα απ' όλα αναφέρθηκε και ο κύριος Ντεμόντ σε αυτό το οποίο είναι το μεγάλο ζήτημα. Και είναι πάρα πολύ απλά απαράδεκτο η διαμάχη μεταξύ δύο κρατών μελών της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για το καθεστώς του Γιβραλτάρ να μπλοκάρει και να έχει όμοιρο ολόκληρο τον ευρωπαϊκό κλάδο της αεροπορίας. Και τι γίνεται. Ευνοούμε τους ανταγωνιστές μας όταν δεν έχουμε έναν ευρωπαϊκό ουρανό, είτε μιλάμε για τα δικαιώματα των επιβατών, είτε μιλάμε για το μπλοκάρισμα που υπάρχει στο Συμβούλιο. Και ακριβώς είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης ε, που εμποδίζει να εκδιπλώσει το δυναμικό του ο ευρωπαϊκός κλάδος αεροπορίας. Δεύτερον, όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούνται πρακτικές ε, σε τρίτες χώρες, στην Τουρκία, στις ε, ε, χώρες του κόλπου και να μην αντιμετωπίζονται καθόλου. Δεν μπορεί να υπάρξει έτσι ανταγωνισμός δίκαιος και θα πρέπει η Κομισιόν να τα πει αυτά ξεκάθαρα στην έκθεση και να δούμε το τι ε, θα γίνει με την αναθεώρηση του κανονισμού 868 ε, του 2006. Και βεβαίως θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον εισηγητή για την ξεκάθαρη έκθεσή του. Αλλά βεβαίως αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι στο σημείωμα ε, κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να μπουν στην ίδια τη γνωμοδότηση. Θα καταθέσουμε οπωσδήποτε κάποιες τροπολογίες, αλλά θα ήθελα να φέρω δύο πράγματα. Σελίδα 10. Μιλάμε για θέμητο ανταγωνισμό, ο οποίος καθορίζεται μέσω γεωγραφικών πλέον εκτιμάτων και ιστορικών ή πολιτισμικών πρακτικών. Μα όταν δεν υπογράφουν τη σύμβαση του ILO οι χώρε του κόλπου. Ε, αυτό δεν είναι κάτι το πολιτισμικό ή ιστορικό. Είναι ένα παράγοντας ανταγωνισμού τον οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Δεύτερον, οι ελεγκτέ εναέρεια κυκλοφορία. Ε, κάμια φορά έχουμε τις απεργίες τους που έχουμε εδώ πέρα στη σελίδες 4 ε, και 5 τα σχετικά, αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθούν ρητός στην έκθεση και τέλος η παρατήρηση που έκανε και ο συνάδελφος ο κ. Κλούνε στην παρατήρηση ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλακεί περισσότερο στην αεροπορία και στις σχετικές συμφωνίες, πρέπει αυτό να μπει στο διατακτικό του κειμένου και όχι μόνο στα εκτιμώντας. Γιατί γνωρίζετε ότι ε, έτσι ε, δεν έχουν το ειδικό βάρος που θα έπρεπε να έχουν. Σας ευχαριστώ. Γκαμπριέλε Πρόης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Νομίζω πως είναι μια καλή βάση για την περαιτέρω συνεργασία μας. Θετικό είναι επίσης το ότι ε, ο εισηγητής ασχολείται με τις συνθήκες εργασίας. Εμείς θεωρούμε πως θα πρέπει να διατηρηθούν, να οι καλές θέσεις εργασίας. Οι αεροπορικές εταιρείες ε, της Ευρώπης ε, δεν χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα δεχτούμε τον αθέμητο ανταγωνισμό μέσω των αεροπορικών εταιρεών του κόλπου. Επιπλέον, Πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ασφάλεια στα αεροδρόμια. Εδώ πέρα ασχολείστε μόνο με την οικονομική πτυχή, αλλά η ασφάλεια στα αεροδρόμια είναι βασική πτυχή και πρέπει να επιμείνουμε σε επαρκώς εκπαιδευμένο και επαρκές προσωπικό. Δεν υπάρχει αυτό στην έκθεση. Το να βασιζόμαστε επίσης τύφλα σε τεχνολογικέ λύσει δεν θα βοηθήσει για να αυξηθεί η ασφάλεια των επιβατών. Επίσης η προκαταγραφή των επιβατών αυτό βεβαίως θα βοηθήσει το κόστος των αεροδρομίων, αλλά εγώ το απορρίπτω. Οι επιβάτες οι οποίοι θέλουν να διαφυλάξουν ιδιωτικότητά τους δεν θα πρέπει να έχουν κάποιο μειονέκτημα. Και βεβαίως θα καταθέσουμε και τις σχετικές μας τροπολογίες όσον αφορά τον κανονισμό της ΕΑΖΑ. Σας ευχαριστώ και είναι Μάισνερ, ναι. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, είναι πολύ καλή η έκθεση. Πόσο σημαντική είναι η αεροπορία νομίζω το είδαμε αυτό γιατί είδαμε ότι το ζήτημα δεν αφορούσε πλέον τις θέσεις εργασίας μόνο αλλά και πάρα πολλούς ε, ανθρώπους στην παραγωγή. Κοιτάξτε, θα αυξηθεί η κίνηση και στον αέρα και παγκοσμίω και πρέπει να βρούμε μια στρατηγική. Αν δεν είναι οι μεταφορές άμεσα από και προς την Ευρώπη, θα χάσουμε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια στρατηγική ανταγωνιστική για το μέλλον. Αυτό ήθελα να πω. Είναι νομίζω πάρα πολύ συναρπαστικό αυτό το οποίο λέμε για το Open Skies. Βλέπουμε πόσες τρελές πτήσεις έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός ουρανός. Και κάτι άλλο να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Εγώ θέλω, πέρα από τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείε και συνδέσεις, να δούμε και το θέμα της γενικής αεροπορίας, ε, των μικρών αεροσκαφών δηλαδή, ε, και των ιδιωτικών αεροσκαφών, γιατί και αυτό αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους και από πλευρά χόμπι, αλλά και από πλευρά απασχόλησης. Και το ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα και εγώ να μιλήσω τώρα στην αεροπορία ε, δεν ε, τίθεται ζήτημα ε, οικονομικής οικονομίας της αγοράς. Ανέφερε και ο κύριος Πρόης, οι αεροπορικές εταιρείε λαμβάνουν 30 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο επιδότηση υπό την έννοια ότι δεν πληρώνουν φόρο στα καύσιμα στην κυροζήνη και αυτό είναι πάρα πολύ άδικο και για λόγους κλιματικούς βεβαίως νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές θα πρέπει να έχουν αεροπορικές συνδέσεις και εκεί πέρα πρέπει να επιδοτούνται. Δεν είναι δυνατόν. Μιλάμε για διασφάλιση της κινητικότητας εκεί, αλλά τώρα να, αυτό δεν γίνεται να ισχύσει για τους πάντες, γιατί παρά τα 30 δισεκατομμύρια αυτά, στην Γερμανία έχουμε πάρα πολλά ε, γύρω στα 23 διεθνή αεροδρόμια, τα 17 είναι ελληματικά. Στην ε, Καναδά όλα τα αεροδρόμια είναι κερδοφόρα γιατί έχουν τόσο ψηλά τέλη. Και ακριβώ εκεί πέρα δεν υπάρχουν εταιρείε low cost γιατί λένε θα πληρώσουν οι επιβάτε το κόστο και τέλο. Δύο παραδείγματα. Στη Γερμανία, στο Κάσελ φτιάξαν ένα καινούριο αεροδρόμιο για 270 εκατομμύρια που είναι μια μισή ώρα από το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Ε, υπάρχουν 3.000 πτήσεις μεταξύ Στουτγάρδης ε, και Φραγκφούρτης, θα μπορούσαν να παίρνουν, το τρένο. <laughs> και τι γίνεται, πέντε αεροδρόμια στην Ρουμανία έχουν 5.000 επιβάτες. Δηλαδή, αντί να επιδοτούνται συνεχώς κάθε χρόνο, το καλύτερο θα ήταν οι χώρες αυτές να έχουν καλύτερους σιδηροδρομικές συνδέσεις Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάμε. Όχι ανάπτυξη με κάθε τίμημα. Μόνο στοχευμένη. Και τώρα ξεχάσαμε την κυρία Ντανιέλα Αγιούτο, η οποία βεβαίως έχει το λόγο. Δεν υπάρχει πρόβλημα κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, συντομία. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την έκθεση, είναι καλή βάση κίνησης. Ήθελα να σταθώ στην παράγραφο 12 σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις. Χαίρομαι διότι υπενθυμίζουμε το ότι οποιαδήποτε χρηματοδότηση, ιδιαίτερα για τα περιφερειακά αεροδρόμια, θα πρέπει να κινείται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Γιατί στα περιφερειακά αεροδρόμια συμβαίνουν πολλά σε ορισμένα κράτη. Δηλαδή υπάρχουν συγκαλυμμένες ε, κρατικές ενισχύσεις, όπου φαίνεται ότι γίνεται διαφορετική χρηματοδότηση από την τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζονται υποστήριξη, αλλά αυτή η υποστήριξη δεν μπορεί να βρίσκεται στις πλάτες των τοπικών φορέων. Θα ήθελα το Κοινοβούλιο να εμπλακεί στην όλη διαδικασία για να βοηθήσουμε και τα περιφερειακά αεροδρόμια που χρειάζονται τη βοήθεια αυτή, γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ορισμένες ευρωπαϊκές ε, περιφέρειες όμως, ε, δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε τις περιφέρειες ή την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί για να κρατήσουν τεχνητά ε, στη ζωή περιφερειακά αεροδρόμια, πρέπει να αφαιρέσουν χρηματοδοτήσεις από άλλους τομείς σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών, θα ήθελα σε αυτό το πλαίσιο να μιλήσουμε για μία φορολόγηση καυσίμων έτσι ώστε να μην μπορούν οι, τα κράτη να αποφύγουν αυτό αυτές, ε, αυτές τις νέες οδούς έτσι ώστε να περάσουν από κράτη που έχουν χαμηλότερα, ε, χαμηλότερη φορολόγηση και να χρησιμοποιούν αυτά τα κράτη. Αυτό δεν επιτρέπεται. Ναι. ναι. Ε, σας θέωσα το λόγο, εντάξει, αλλά μακρηγορήσατε λίγο. Λοιπόν, για την Κομισιόν τώρα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που επανήλθα στον κόσμο της αεροπορίας και χαίρομαι για τα όσα έγιναν εν τη απουσία μου και χαίρομαι που ξανά ήρθα στην Επιτροπή. Ευχαριστώ μου δώστε το λόγο. Καλώς ήρθατε λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Επίσης να ξεκινήσω με κάτι θετικό. Να συγχαρώ τον κύριο Ταλίτσκα για την εξαιρετική έκθεση για την στρατηγική για την αεροπορία και να κάνω κάποια σχόλια εκεί όπου είναι η θέση της Κομισιόν να Συμφωνώ με τον κύριο Τελίτσκα για την έμφαση που δίνει στην συνδεσιμότητα. Σαφώς ε, πρώτε, η προτεραιότητα για όλους μας. Έχει σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία και πολλοί ήδη το είπαν ότι η συνδεσιμότητα βεβαίως ε, είναι άνηση και αυτό οδηγεί σε κάποια μειονεκτήματα. Οπότε συμφωνούμε πλήρως με αυτό. Επίσης συμφωνούμε με το βάρος που δίνεται στην ασφάλεια της αεροπορίας. Όσον αφορά τώρα τους διάσημους αυτοκινητοδρόμους των εθέρων και τον κανονισμό 351, συμφωνούμε ότι είναι κάτι το πολύ ενδιαφέρον και ζητήσαμε τον διαχειριστή του δικτύου να κάνει μια μελέτη, να δούμε δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον εναέριο χώρο της Ευρώπης και ένα μέσο για να πάμε προς το νέο ευρωπαϊκό ουρανό. Φοβάμαι ότι τίποτα δεν έχει προχωρήσει στον τομέα αυτόν και είναι απογοητευτικό το ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδο. Ελπίζουμε η μελέτη σκοπιμότητας να καταστήσει σαφή τα ωφέλη και το κόστο για να τα δούμε όλα προσεκτικά. Η κυρία Κλούν τόνισε την σημασία των συμφωνιών των αεροπορικών και σα ευχαριστώ για τη στήριξή σα. Και αν μου επιτρέπετε, ε, νομίζουμε πω έχετε δίκιο στόχο έχουμε ακριβώς ε, να είμαστε σε επαφή με τις αναψώμενες περιοχές του κόσμου για να έχουμε και εμείς ανάπτυξη για δουλειές αναφέρατε τον δείκτη συνδεσιμότητας συγκεκριμένα. Αυτό έπρεπε να το έχω πει πριν. Μετά από συνεργασία με το Eurocontrol μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε ακριβώς όλες τις υφιστάμενες ε, ρυθμίσεις με βάση αυτά Προς την κυρία Γιάλα και την κυρία Πρόισον αναφέρατε και οι δύο την σημασία του κοινωνικού διαλόγου. Συμφωνούμε επ' αυτού. Βεβαίω το θέμα του εργατικού δικαίου και, και η επιβολή του είναι θέμα των κρατών μελών, αλλά προσπαθούμε πάλι ακριβώ να στηρίξουμε τον κοινωνικό διάλογο μέσω του της Κλαδικής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου για την Πολιτική Αεροπορία, και βέβαια να δούμε το θέμα της απασχόλησης και βέβαια να μένουμε τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών. Κάποιοι ανέφεραν τα δικαιώματα των επιβατών. Ναι, συμφωνούμε για την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος. Ο κανονισμός είναι πάνω από 10 ετών. Έχει υπάρξει υπερβολική ερμηνεία και περιμένοντας την νομοθεσία η οποία δυστυχώς έχει μπλοκαριστεί εκδώσαμε αυτές τις ε, ερμηνευτικές εγκυκλίους, οι οποίες βεβαίως πλέον ε, όταν τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός θα είναι παροχημένες, αλλά ακριβώς σκοπεύουμε να βρούμε την ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων των επιβατών και του οικονομικού κόστους αυτών. Κάποια άλλα ενδιαφέροντα σχόλια αφορούσαν ακριβώς το πρόβλημα δυναμικότητας των αεροδρομίων που είναι πλέον ζήτημα και ελπίζουμε κάποια πράγματα που έχουν μπλοκάρει, ο ενιαίος ουρανός 2 ε, και ο κανονισμός περί χρονοθυρίδων να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Τέλος, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και τα αεροδρόμια στο παρατηρητήριο των αεροδρομίων και ελπίζουμε να έχουμε κάποιες βέλτιστες πρακτικές οι οποίες θα εφαρμοστούν όσον αφορά το σχεδιασμό των αεροδρομίων. Εάν τώρα μου επιτρέπετε να επανέλθω στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε η κυρία Φώστερ και ευχαριστούμε για την σταθερή στήριξή της στο θέμα αυτό. Τώρα, υπήρχε ένα άλλο σχόλιο για τα κοινωνικά. Α, συγγνώμη. Δεν βλέπουμε λοιπόν στοιχεία μέχρι στιγμής πως τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα ε, επιδρούν στα ζητήματα ασφαλείας. Είναι ένα σημαντικό θέμα και είναι γεγονός πως οι πολυεθνικές εταιρείες δύσκολα υποπτεύονται από τις εθνικές αρχές, οπότε προσπαθούμε να δούμε πώς θα ενισχύσουμε την δυνατότητα εποπτείας των πολυεθνικών εταιριών που έχουν βάσεις διασπαρμένες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα μπορούσαμε ακριβώς να μοιράσουμε τις δυνατότητες των κρατών μελών μεταξύ αυτών και της ΕΑΖΑ. Οι κύριοι Ντεμόντε και Βαν Χίλτενμπεργκ ανέφεραν και οι δύο βεβαίω ε, το... τον ελέφαντα στο δωμάτιο, τον βράχο θα έλεγα εγώ, το Γιβραλτάρ. Συμφωνώ πλήρω. Πολλά ζητήματα τη αεροπορία έχουν κολλήσει. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Και εμεί συζητάμε και από τι δύο πλευρές να επιδείξουν ένα επικοδομητικό πνεύμα Νομίζω πως δεν είμαι ο πρώτος από την Κομισιόν που το λέει αυτό. Ναι. Για το θέμα των περιφερειακών αεροδρομίων και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Θεωρούμε πως οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που εγκρίναμε το 2014 είναι σημαντικό ζήτημα για την σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και βεβαίως ελπίζω έτσι να έχουμε μια καλύτερη αίσθηση των προκλήσεων των περιφερειακών αεροδρομίων. Έγινε διαβούλευση εξαντλητική. Νομίζουμε ότι καταφέραμε να λάβουμε υπόψη τις αλλαγές στην αγορά της τελευταίας δεκαετίας ε, με τις προτάσεις μας. Ελπίζω λοιπόν να έκανα κάποια σχόλια τα οποία θα σας βοηθήσουν στην έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και χαίρομαι που επανήλθα στην Επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ. Είναι λοιπόν ξανά η πρώτη φορά. Οπότε τον λόγο έχει ο κύριος Τέλιτσκα. Uh, Συνάδελφοι, νομίζω ότι εσείς ε, έχετε συντάξει πολύ καλύτερες εκθέσεις από εμένα, γιατί εγώ βρίσκομαι στο Κοινοβούλιο όχι για μακρύ διάστημα όπως γνωρίζετε γι' αυτό. Ε, θα ήθελα, όπως είπε ο κύριος Βαντερκάμπ, να με συμπεριλάβουμε θέματα τα οποία δεν έχουν ε, συμπεριληφθεί και θα ήθελα αυτό να αντικατοπτρίζεται και από τις δικές μου τροπολογίες. Στην αιτιολογική έκθεση βλέπετε ποιες είναι οι προθέσεις μου. Μίλησα και για τις συμφωνίες αερομεταφορέων, και αυτό το βλέπετε και στην έκθεση. Στην έκθεση καλούμε τον Επίτροπο να ε, ασχοληθεί με θέματα στα οποία αναφερθήκατε κι εσείς, μιλήσατε για χρονοθυρίδες, για τους ελεγκτές κυκλοφορίας και ούτω καθεξής. Πάση περιπτώσει, Υπάρχει θέμα εφαρμογής, δηλαδή έγινε πρόοδος, αλλά δεν ε, εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές όπως θα έπρεπε. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ξεμπλοκάρουν αυτή την κατάσταση για να στείλουμε και ένα μήνυμα από πλευράς Ευρωκοινοβουλίου. Μιλήσατε για περιφερειακά αεροδρόμια από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Πιστεύω ότι στόχος είναι η οικονομική βιωσιμότητα, δηλαδή να μην κάνουμε επενδύσεις σε μια οδό η οποία, οι οποίες θα χαθούν. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε δύο ή τρία αεροδρόμια μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, ολοκλήρωσης, αλλά αν υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση που θα σας ε, οδηγήσει να φτάσετε πολύ νωρίτερα, τότε θα πρέπει να επενδύσουμε στα τρένα. Μίλησατε για την πολιτική ανταγωνισμού. Θα πρέπει να πω ότι δεν είναι εύκολο το όλο ζήτημα. Αν όμως υπάρχει ζήτηση από τους επιβάτες, τότε αυτό είναι κάτι που μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη. Μπορούν να το προσφέρουν οι αερομεταφορείς έτσι ώστε να μην χάσουμε επιβάτες. Αν χάνουμε επιβάτες θα πρέπει να δούμε γιατί. Αν κάποιος ε, ε, δρά με αθέμητο ανταγωνισμό, που θα πρέπει να δράσει η Επιτροπή και όπως ε, γνωρίζω έχουν γίνει, έχει γίνει προσφυγή από πολλούς, ε, από πολλούς. Γιατί δεν υπάρχει λοιπόν συμμόρφωση. Υπάρχει προστατευτισμός, υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Ή θα πρέπει να δούμε τη χρήση αυτών των προτύπων. Αυτό θα με απασχολήσει αλλά ίσως να μην σας ικανοποιήσω όλους γιατί εγώ δεν θα σταθώ υπέρ του προστατευτισμού και κατά των Ευρωπαίων καταναλωτών και επιχειρήσεων. Έχω καταγράψει όλα τα σχόλια, μπορεί να μην αναφερθώ βέβαια σε όλα τώρα. Το περιβάλλον είναι κάτι που θα με απασχολήσει λεπτομερώς ένα ε, ε, ε, ζήτημα αφορά την κυκλική οικονομία. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε με πολλές δυνατότητες, μία νέα δυναμική σε αυτό το τομέα και μπορούμε να δούμε τι γίνεται στα αεροδρόμια, τι γίνεται μεταξύ αεροδρομίων, ποια είναι η συνδεσιμότητα και ούτω καθεξής. Θα σταματήσω εδώ γιατί μας πιέζει ο χρόνος, αλλά πιστεύω ότι ασχολήθηκα με τα περισσότερα σχόλια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, Σκιώδης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήμουνα σε σταθερή επαφή με την Κομισιόν και θα ήθελα να πω ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά από εμάς σε σχέση με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ή την επιτυχία. Ως προς το κοινωνικό καθεστώς, το, το κοινωνικό τομέα θα πρέπει να δούμε το θέμα από πλευράς μεταφορών. Είμαστε η Επιτροπή ε, Τραν. Ε, νομίζω όμως ότι δεν θα πρέπει να αντικαθιστούμε άλλες επιτροπές στο έργο τους. Ο Πρόεδρος Κράμερ, ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών είναι 5η δεκάτου στις 12 το μεσημέρι. Τώρα Είμαστε καλά από, από ψυχρόνου θα έλεγα. Ερχόμαστε στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Η συγκήτρια η κυρία Μάισνερ. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε κάποιο χρόνο. Βέβαια το θέμα της ναυσιπλοείας είναι πολύ σημαντικό. Είπα πριν και για την aviation ότι βεβαίω οι μεταφορές θα αυξηθούν. Το ίδιο και στην εσωτερική ναυσιπλοεία που μπορεί να ε, μεταφέρει μια στιγμή διακόπτη πρόεδρος. Σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία και εφόσον επιθυμείτε να εξέλθετε, να εξέλθετε με ησυχία. Δεν είναι δυνατόν να ενοχλείτε, η κυρία Μάσινερ την ώρα που ομιλεί από το θόρυβο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν ότι οι οδοί της εσωτερικής ναυσιπλοείας πρέπει να επεκταθούν διότι μπορούν να ε, βοηθήσουν πολύ στο μεταφορικό έργο και να ξαλαφρώσουν και το δρόμο. Για να γίνει αυτό όμως χρειαζόμαστε ανθρώπους με εκπαίδευση και κατάρτιση. Ήδη υπάρχει πρόβλημα. Τα πληρώματα των σκαφών που κινούνται στην εσωτερική ναυσιπλοεία είναι ήδη γερασμένα και δεν υπάρχουν αντικαταστάτες. Ούτε σχετική εκπαίδευση. Θα ήταν σωστό να γίνει μια πρόταση εναρμόνισης για την κατάρτισή τους. Ομολογώ ότι έμαθα πολλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζω ότι για παράδειγμα στη Φιλανδία υπάρχουν επιπλέουσες σάουνες που δεν είναι ακριβώς βεβαίως ε, σκάφος ε, με την έννοια του σκάφους που εκτελεί εσωτερική ναυσιπλοεία αλλά είναι ε, επιπλέον, είναι πλωτά μέσα. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι δύσκολο να συνταχθεί τέτοια έκθεση για το Κοινοβούλιο όταν το Συμβούλιο έχει ήδη κάνει τη δουλειά του, έχει ήδη τελειώσει τα μαθήματά του, έχει ήδη κάνει την εκθεσή του. Εγώ θα έρθω λοιπόν τώρα στα διάφορα επιμέρους θέματα όπου ζητώ κάποιες τροποποίησεις. Γενικώ δηλαδή είναι σωστό να προτείνεται η εναρμόνιση. Άλλωστε είναι και κάτι που εξυπηρετεί την κινητικότητα για την εκπαίδευση. Επειδή είμαι από το Μέκλεμπουργκ, ε, Δυτική Πομερανία, όπου ε, χρειαζόταν να γίνουν ε, σχετικές διατάξεις, Εκεί είχαμε και ένα θέμα με ε, τους... Ε, με ε, ε, ένα ειδικό είδος μεταφοράς. Λοιπόν, χρειάστηκαν ειδικέ διατάξεις. Ε, τώρα, εμείς εδώ, αυτά δεν ισχύουν βέβαια για όλη την Ευρώπη. Εδώ χρειάζονται και να δημιουργηθούν κάποιες σχολές που θα εξυπηρετούν την ανάγκη αυτή. Και υπάρχουν και ορισμένα ε, ζητήματα όπου ζητεί απελευθέρωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπε για παράδειγμα ότι όταν δεν διασυνδέονται με άλλες εσωτερικέ αυτές οδοί ναυσιπλοείας, τότε μπορούν να εξαιρεθούν. Ε, εγώ γνωρίζω ότι στη Γερμανία τα πολύ μικρά οχήματα αγωγά μπορούν όντω να εξαιρεθούν από την ανάγκη εκπαίδευση του προσωπικού, αυτό εννοώ του πληρώματο δηλαδή, και σε πολύ μικρέ διαδρομέ. Η γνώση των διαδρομών επίσης είναι πολύ ε, σημαντικό να περιληφθεί στα προγράμματα διδασκαλίας, δηλαδή που έχουν οι διάφοροι ποταμοί ε, κάποιες δυσκολίες, αβαθή κλπ. Εγώ βλέπω ως κριτήριο ότι έχουν αυξηθεί τα ναυτικά ατυχήματα σε ορισμένα σημεία ποταμών. Και θα πρέπει να εξετάζεται ο εκπαιδευόμενος και αν έχει τη σχετική γνώση. Βεβαίω είναι διαφορετικοί οι διάφοροι ποταμοί που εξυπηρετούν την εσωτερική ναυσιπλοή και σε ό,τι αφορά τα ρεύματά του κλπ. Η αναγνώριση τρίτων χωρών τώρα εκεί εφόσον η τρίτη χώρα έχει διασύνδεση με εσωτερικών ε, οδών ναυσιπλοείας και με χώρε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε ναι. Αν όμω είναι αλλού στον κόσμο πώ θα εξετάσουμε τώρα εάν οι τρίτε χώρε αυτέ. Ε, σέβονται τα όσα γράφουμε εμείς εδώ. Οι εξετάσεις μπορούν να γίνονται και σε simulator, σε απεικονιστή. Μπορούν, α, ε, μπορεί με τον τρόπο αυτό να παιχθούν εντό εισαγωγικών και ε, πολύ δύσκολα σενάρια, τα οποία είναι πολύ δύσκολο βέβαια να εξεταστούν στην πράξη. Βέβαια, το simulator δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πράξη πράγματι ε, ε, στο ποτάμι. Υπάρχει και η οργάνωση ΣΕΣΝΗ που έχει ε, ήδη θεσπίσει προδιαγραφές και θα είναι σωστό να τις λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλοι οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές ειδικότητες, εάν δεν υπάρχουν επαρκείς καταρτιζόμενοι, θα πρέπει να είναι δυνατόν να προσέλθουν από άλλη ε, ειδικότητα, από άλλο κλάδο. Ίσως ε, συγγενή κλάδο δηλαδή, από τις θαλάσσιες μεταφορές για παράδειγμα. Αυτό είναι θετικό και ορθό βρίσκω κατά τα λοιπά, προβαίνω σε συμπλήρωση. Ο επικεφαλής, ο πλοίαρχος ας πούμε, θα πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι δραστηριότητες που διεξάγονται επί του σκάφους. Υπάρχουν για παράδειγμα πολύ μικρά πληρώματα. Κάποιο ο οποίος διευθύνει το πλοίο θα πρέπει να γνωρίζει όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες ώστε εν ανάγκη να μπορεί και αυτός να κάνει κάτι. Τέλος, είμαι υπέρ των Αγγλικών στην περίπτωση αυτή. Και με τον τρόπο αυτό θα δει να περιθούν και τα αγγλικά στο ορολόγιο πρόγραμμα. Οι σκιώδεις είμαι υποχρεωμένος να σας περιορίζω το χρόνο σας στα δύο λεπτά. Ενώ Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ποιότητα αυτής της έκθεσης. Το ΕΛΚ είναι πεπισμένο ότι η προσέγγιση της Κομισιόν είναι πολύ καλή για τον επαγγελματισμό σε αυτό το τομέα. Επίσης θα πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένα πρότυπα και προδιαγραφές για την εσωτερική ε, ναυσιπλοεία. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις για τις εσωτερικές πλωτές οδούς που δεν συνδέονται με το ευρωπαϊκό δίκτυο. Και επίσης να μιλήσουμε για μία ενδεχόμενη συμφωνία Επίσης, το πλαίσιο αυτό δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για τους επαγγελματίες. Θα πρέπει τα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν όπως ορίζονται στα παραρτήματα. Ξεκινάμε πολύ καλά και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει συμφωνία αν παραμείνουμε στα τρία αυτά σημεία. τα Ταπαντέλ και σας παρακαλώ να είστε και σύντομοι. Λοιπόν, τα Ταπαντέλ. Το γοργόν και να έχει, ε. Λοιπόν, ε. λοιπόν Κλαούντια Ταπαντέλ μικρόφωνο. Αγαπητοί συνάδελφοι, Γκεζίν, θα ήθελα να, σα, να σε ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική για τον ε, τομέα των ε, μεταφορών. Θα βοηθήσει και για το εργατικό δυναμικό. Είναι ισορροπημένη η έκθεση σε σχέση με τα επαγγελματικά προσόντα καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να λύσουμε το θέμα των αρμοδιοτήτων. Θα ήθελα να ε, αναφερθώ σε αυτά που είπε η Γκεζίνε. Σε σχέση με την ψηφιοποίηση, η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει, μπορεί να γίνονται πολύ πιο γρήγορα επαληθεύσεις και να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων και να μειώσουμε και την ε, γραφειοκρατία σε σχέση με το, τον προσωμιωτή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ε, υποκαταστήσει την πραγματική εργασία. Νομίζω ότι η πραγματική δράση, ιδιαίτερα όταν είμαστε υπό στρες, οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Γι' αυτό ένας προσωμιωτής δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να υπάρχει η σωστή προπαρασκευή σε σχέση με την πιστοποίηση και ε, αναφέρομαι στον αριθμό ημερών, βλέπουμε ότι παρατάθηκε αυτή η προθεσμία. Δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να παραταθεί, να γίνει αυτή η παράταση, παράταση βεβαίως. Μπορούμε να το συζητήσουμε με την Κεζίνε. Ένα βασικό θέμα αφορά τις ζώνες κινδύνου. Θα πρέπει να ορίσουμε αυτές τις ζώνες για να μειώσουμε τους κινδύνους, έτσι ώστε να μην ενταχθούν βρεθούν αυτές οι ζώνες σε αυτή την κατηγορία επικινδυνότητας. Τα κράτη-μέλη μπορούν να ορίσουν αυτές τις ζώνες, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η έκθεση είναι πολύ σημαντική, γι' αυτό δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να περιοριστεί σε ένα-ενάμιση λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτό πρέπει να τηρήσουν όλοι τον χρόνο. Λοιπόν, Πέντερ Φαντάλεν, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πως ε, η Κομισιόν έχει κάνει μια καλή πρόταση να το υπογραμμίσω. Δεύτερον, και η κυρία Μαϊστινέρε έχει κάνει κάποιες καλές συμπληρώσεις στην εκθεσή της για τα επεγγελματικά προσόντα των κυβερνητών που θα πρέπει να, είναι, να έχουν μακροχρόνια ισχύ και βέβαια για τη χρήση των αγγλικών στην ιστορική ναυσιπλοεία. Υπάρχει στην ναυτιλία την πόρο το λεγόμενο c Speak, ε, ένα λεξιλόγιο που μπορούν να συνεννοούνται οι άνθρωποι. Κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχει και Βεβαίω στην εσωτερική ναυσιπλοή, γιατί ε, συχνά έχουμε κάτι ναύτες οι οποίοι μιλάνε κάτι ε, λίγα αγγλικά και αυτή τη γλώσσα θα γνωρίζουν όλοι. Επίσης Πρέπει να δούμε τα ζητήματα των ορισμών ε, πάρα πολύ προσεκτικά. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ε, πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση το θέμα. Ευχαριστώ που τηρήσετε και τον χρόνο. Μαρία Κελνέν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Μάισνερ για την επαγγελματική έκθεση και βεβαίως την Κομισιόν. Εμείς έχουμε προτείνουμε κάποιες αλλαγές στο κείμενο αλλά θα έλεγα ότι ως φίλοι των, ε, της εσωτερικής ναυσιπλοείας θα ήθελα να υπάρχει και στο μέλλον και να υπάρχει και μια συνέχεια, λαμβάνοντα υπόψη ότι όσοι εργάζονται σε αυτόν τον κλάδο δεν είναι μια ενιαία ομάδα. Ε, είναι διαφορετικοί άνθρωποι που δουλεύουν από διαφορετικές ε, συνθήκες από μικρές ε, εταιρείες μέχρι πολυεθνικές και βέβαια και ασφάλεια είναι το βασικό ζήτημα. Όμως, χωρίς βεβαίως να προκαλούμε αξεπέραστα διοικητικά βάρη στις ε, μικρές εταιρείες έτσι ώστε να μην μπορούν πια να λειτουργούν. Θεωρώ πως η εσωτερική ναυσιπλοεία στο μέλλον θα είναι πάρα πολύ σημαντική και στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και των επιβατικών και είναι σημαντικό για να μειωθούν και οι κομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ. Μαρίν Κριστίν Νοτιού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ τον κύριο Θεολογίτη και τους συναδέλφους του που προσήλθαν για να μας μιλήσουν για αυτή την πρόταση οδηγίας. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση για τη... την ένταξη αυτή του επαγγέλματος και τον προσδιορισμό του ως προς τις ε, εσωτερικές πλωτές οδούς. Όπως ξέρετε, εμείς γνωρίζουμε μεγάλα προβλήματα στο τομέα της ναυσιπλοείας. Είχαμε 10.000 ε, επλοία και τώρα ε, έχουμε πάρα πολύ λιγότερα, κάτω από τα χίλια. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους ε, πλειοκτήτες, γιατί υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε έναν Γάλλο ο οποίος θα ε, πλέψει στο Δούναβι σε σχέση με έναν Ρουμάνο ο οποίος θα χρησιμοποιήσει το, τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Γαλλίας. Αυτό ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί το θέμα των αρμοδιοτήτων είναι πολύ καλό, αλλά θα πρέπει να δούμε και αυτά τα επιμέρους σημεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που επένεσαν την κυρία Μάισνερ. Συμφωνώ λοιπόν και εγώ. Έχω δύο ερωτήσεις. Θα έχουμε τώρα ένα ευρωπαϊκό σύστημα προσόντων για την εσωτερική ναυσιπλογία, ναι ή όχι η Κομισιόν έχει κατεβάσει μια πρόταση έτσι και έτσι. Είτε να συντονιστούν τα εθνικά συστήματα ή θα έχουμε άλλα συστήματα. Τι θα κάνουμε. Δεύτερη ερώτηση. Αν απαιτείται μακροχρόνια εμπειρία, λένε καμιά φορά 500 μέρες και δεν ολοκληρώνεται με κάποια εξέταση, δεν ξέρουμε αν ε, γνωρίζει κάποιος το αντικείμενο. Είτε μικρότερη περίοδος με εξετάσεις ή μεγαλύτερη περίοδος χωρίς εξετάσεις. Αν θα μπορούσατε να απαντήσετε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω και άτομα με διπλώματα που δεν έχουν ιδέα και άτομα χωρίς διπλώματα που δεν ξέρουν τη δουλειά. Αλλά βεβαίως η ερώτηση είναι προς την Κομισιόν. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον κύριο Θεολογίτη. Ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Θα ήθελα με τη σειρά μου να συγχαρώ την εισηγήτρια κυρία Μάισνερ για την θαυμάσια έκθεση που έχει συντάξει. Με χαρά είδαμε ότι όχι μόνο η εισηγήτρια αλλά και οι άλλοι ευρωβουλευτές που παρενέβησαν τοποθετήθηκαν θετικά υπέρ της προτάσεως, διακρίνουν την προστιθέμενη αξία της ό,τι αφορά την ασφάλεια και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, πράγμα που χρειαζόμαστε για να προωθήσουμε περισσότερο αυτή την φιλική προς το περιβάλλον υπηρεσία που προσφέρει η εσωτερική ναυσιπλοεία. Έχουμε κάποι... Ε, έχετε κάποια σχόλια μάλλον, δεν θα τα ε, σχολιάσω διαμακρών. Ε, ερώτηση της αξιολόγησης Δηλαδή, αν θα αφοργείται πιστοποιητικό χωρίς αξιολόγηση, αυτό όμως θα υποσκάψει ολόκληρη την ε, προσέγγιση. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, εάν περιορίσουμε τον αριθμό των προσώπων, η λειτουργούσα ενιαία αγορά θα περιοριστεί πάρα πολύ. Ε, από άποψη τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς δηλαδή στην περίπτωση αυτή, θα περιοριστεί πάρα πολύ. Ούτε μας αρέσουν πολύ οι εξαιρέσει που όλο και περισσότερες εξαιρέσει θα οδηγήσουν τελικά σε ένα κατακαιρματισμό των εθνικών περιπτώσεων. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει μια ενιαία, πραγματικά ενιαία αγορά. Μια ενιαία σφραγίδα για μια ενιαία αγορά. Στην προσπάθειά μας για εξασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερο γραφειοκρατικό άχθος και εμπόδια για την είσοδο στο επάγγελμα, όπως είπαν κάποιοι από τους παρεμβάντες για τις διαδρομές που έχουν ιδιαίτερους κινδύνους. Βεβαίως υπάρχουν ποτάμια που έχουν ιδιαίτερους κινδύνους, αλλά το επιχείρημα αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να περιοριστεί τεχνητά η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Τέλος, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές πτυχές της προτάσεως, εάν δηλαδή θα διευκολύνει με κάποιον τρόπο την ένταξη προσώπων που δεν θα εργάζονται υπό τις ίδιες συνθήκες και επομένω θα πετάξουν έξω από την αγορά κάποιους άλλους. Αυτό βεβαίω η πρότασή μα δεν θα είναι η λύση όλων των κοινωνικών προβλημάτων στι μεταφορέ, ασφαλώ όχι, αλλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε εδώ είναι να μην επιτρέψουμε ένταξη στην αγορά αυτή εργασία προσώπων χωρί την απαραίτητη κατάρτιση. Ήδη αυτό θα ανεβάσει το επίπεδο, γιατί δεν μιλούμε μόνο για του boat masters, αλλά για όλα τα επίπεδα τη εκπαιδεύσεω. Εν τέλει, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι όπως πάντοτε θα συνεργαστούμε επικοδομητικά μαζί σας για να φτάσουμε στην καλύτερη δυνατή ισορροπία για την διευκόλυνση της εσωτερικής ναυσιπλοείας, την εξασφάλιση υψηλού επίπεδου ασφαλείας. Και αν μου επιτρέπετε να καταχαστώ για λίγο τον χρόνο σας, γνωρίζω κύριε Πρόεδρε ότι, ότι ε, βιάζεστε, δώστε μου ένα λεπτό για να κάνω μια προσωπική παρατήρηση. Είναι η τελευταία μου εμφάνιση ενώπιον σας σας έχω συνεδεύσει τα τελευταία 16 χρόνια, από το 2000. Βλέπω μερικούς ευρωβουλευτές οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται εδώ και μου θυμίζουν πάρα πολύ ευχάριστη στιγμές συνεργασίας μαζί σας, είτε για την ε, οδική ασφάλεια, είτε για την ασφάλεια στην αυτιλία, για τα λιμάνια, για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Νομίζω ότι συμβαδίσαμε, συμπορευθήκαμε για ένα μεγάλο διάστημα και σας ευχαριστώ για τη θαυμασία συνεργασία και για την πολύ πάντα επικοδομητική σας στάση απέναντι στις προτάσεις της Κομισιόν. Από τα μέσα Οκτωβρίου θα ε, συνεργάζεται με την Τανιέλα Ρόσκα, η οποία αναλαμβάνει, μιας και εγώ συνταξιοδοτούμε αρχές του επόμενου έτους. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι, καλή συνέχεια και ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμούμε να συνεργαστούμε μαζί σας, μαζί μου είτε στο πρόσωπο της διαδόχου μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ευχαριστώ σας δίαθεσα αυτό το έξτρα λεπτό και είδατε και τα χειροκροτήματα των συναδέλφων μου. Σας ευχαριστώ πάντως και πάλι και προσωπικά όλους ιδιαίτερος και πολύ εγκάρδια για την συνεργασία σας βεβαίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό της αλλά και με εσάς ως πρόσωπο διότι οι θεσμοί τι είναι εάν τα πρόσωπα που τους απαρτίζουν δεν δίνουν το χέρι συνεργασίας. Για την νέα φάση της προσωπικής σας ζωής σας εύχομαι κάθε επιτυχία και μην περιμένετε και πολύ ησυχία στη νέα αυτή φάση της ζωής σας. Και από μένα, κύριε Θεολογίτη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ νομίζω ότι τον Οκτώβριο θα σας ξαναδούμε. Ε, κρίμα. Φαίνεται πως είναι πράγματι τελευταία σας εμφάνιση εδώ. Ε, ε, σας έχω εκτιμήσει όλους ιδιαίτερος πάντοτε και τη συνεργασία μαζί σας, διότι έχω αντιληφθεί ότι είστε κάποιος εκπρόσωπος της Κομισιόν που γνωρίζει για ποιο πράγμα μιλεί. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουν. Ναι, αλλά κάπω έτσι ακούστηκε. Ναι, ναι, γι' αυτό διορθώνω την εντύπωση αυτή. Αλλά εγώ έχω, ασχολούμαι πολύ με τα λιμάνια. Κάθε φορά που πήγα, ε, εγώ είμαι από το Αμβούργο, και κάθε φορά που πάω εκεί να του συζητήσω ένα θέμα, μου λένε Α, μόλι πριν από μια εβδομάδα ήταν εδώ ο θεολογήτη ή θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Άρα δεν είναι άνθρωπο ο οποίο ε, κάθεται στο γραφείο του και σκέφτεται πράγματα, αλλά πηγαίνει επιτόπου και ασχολείται. Γι' αυτό λοιπόν και έχω ε, ασχοληθεί και με πολλά δοσία τα οποία ήταν τη δική σα ευθύνη και βεβαίω έχω πάει και εγώ και έχω δει τον κόσμο επί τόπου και πολύ καλά έχετε κάνει το ίδιο και εσεί. Γι' αυτό χάρηκα πολύ που μπόρεσα να συνεργαστώ μαζί σα, έστω και αν διαφωνούσαμε κιόλα, ε, αλλά και αυτό σημαίνει δημοκρατία. Πολύ σύντομα τώρα για τα όσα λέχθηκαν ήδη μέχρι τώρα στην συζήτηση, που ήταν ακριβώ και τα ζητήματα εκείνα που έχουν κάποια αγκάθια, α το πούμε έτσι. Η οργανωσία για παράδειγμα, περισσότερο θεωρώ εγώ να παίξει ρόλο από ότι η Κομισιόν, ότι δεν χρειάζεται παραπάνω φραγμή από ότι ε, υπάρχουν. Ψηφιο, ψηφιοποίηση θα ήθελα ήδη από τώρα. Simulators δεν μπορούν να αντικαταστήσουν βέβαια την εξέταση στην πράξη. Και αυτό σωστό. Νομίζω ότι υπάρχουν και ορισμένα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε ακόμη για να δούμε τι ακριβώς θα εγγράψουμε ακόμα στην ονομοδότησή μας. Είπατε επίσης, ε, μια συνάδελφός μας, ότι δεν είναι ομοιογενής η ομάδα στην εσωτερική ναυσιπλοεία των, των, ε, των προσώπων δηλαδή που ασχολούνται βεβαίω. Είναι και πολύ διαφορετικά τα μεγέθη των πληρωμάτων και είναι οι διαφορετικέ επιτόπου συνθήκε τη εσωτερική ναυσιπλοεία. Δεν μπορεί λοιπόν να τα βάλει κανεί όλα στο ίδιο κανάθι. Πρέπει να δούμε πώ θα εναρμονίσουμε και σε ποιο βαθμό, λαμβάνοντα ωστόσο υπόψη τι ανάγκε όλων των επαγγελματικών ομάδων. Τέλο. κάθε ένας θα πρέπει να αντιμετωπίζει εξετάσεις. Ε, βεβαίως ε, συμφωνώ, με, θα πρέπει να έχει το πτυχίο δηλαδή από τις εξετάσεις. Ε, βεβαίως συμφωνώ με τον πρόεδρο που είπε ότι μερικοί έχουν δίπλωμα και δεν ξέρουν τίποτα. Και άλλοι ξέρουν πολλά πράγματα αλλά δεν έχουν δίπλωμα. Το θέμα πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον και βεβαίως τέλος η Κλάουδια έχει δίκιο το επειδή αντιμετωπίζουμε πρόβλημα χρόνου να κάνουμε συντομότερες τις Τη ε, οδούς της Ναυσιπλόγια δεν είναι σωστό. Έχετε δίκιο, βεβαίως. Γνωρίζουμε ότι είσαι και η γεννημένη εισηγήτρια για το θέμα αυτό. Τώρα, 11 Οκτωβρίου στις 2 το απόγευμα, η προθεσμία κατάθεσης των τροπολογιών. Και το επόμενο θέμα, οι κανόνες αστικού δικαίου σχετικά με την ρομποτική. Με εισηγητή τον Γεώργιο Μάιερ, ο οποίος όμως αντικαθίσταται σήμερα λόγω απουσίας από την κυρία Αρνοτού. Ο κύριος Μάιερ ζητά συγγνώμη γιατί ε, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, γι' αυτό θα παρουσιάσω εγώ την έκθεση αυτή για το αστικό δίκαιο ε, και τη ρομποτική. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ε, φτιάχνουμε ρομπότ αυτόνομα και ευφυή σε διάδραση με το περιβάλλον και που μπορούν να λάβουν αποφάσεις ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Αυτή η επανάσταση όμως που είναι ε, πραγματικότητα και όχι επιστημονική φαντασία όπως έλεγε ο Ασίμοφ δημιουργεί νομικά και δεοντολογικά προβλήματα. Αυτό που έχει σημασία είναι να βρούμε την προστιθέμενη αξία και την κατανομή της στον τομέα των ε, μεταφορών. Έχει σημασία λοιπόν με βάση την, ε, την, ε, τις πολυτροπικές μεταφορές να δούμε πώς μπορούν να αυξηθεί, να αυξηθεί το κέρδος και στις οδικές μεταφορές, ναυσιπλοεία και ούτω καθεξής. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο καταναλωτής και αυτός που ορίζει το έργο να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο κέρδος. Δηλαδή αυτό μέσα στα πλαίσια μια συγκεκριμένης δράσης και όχι αδράνειας. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς ιδιαίτερα είναι το θέμα των ατυχημάτων. Όταν το όχημα βρίσκεται σε αυτόματο πιλότο και να δούμε ποια είναι τα δεοντολογικά ζητήματα. Βλέπουμε ότι τα οδικά δυστυχήματα θέτουν μεγαλύτερα προβλήματα με βάση τη ρομποτική, αν και έχουν μειωθεί. Παρόλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι η μηχανή είναι πιο αξιόπιστη από τον άνθρωπο. Η Uber μαζί με τη Volvo έκανε τα πρώτα πειράματα χωρίς οδηγό στις ΗΠΑ μέσα στα πλαίσια της αυτοματοποίησης. Αυτό το κάνει και η Google με τη σειρά της. Δεν ε, πρόκειται για θεωρητικές υποθέσεις, αλλά προτρέχουμε ως προς την πραγματικότητα σε ευρεία κλίμακα. Βλέπουμε ότι ήδη έχουν υπάρξει δυστυχήματα. Ποιος είναι υπεύθυνο ο ιδιοκτήτης, ο κατασκευαστής ή τα ρομπότ αυτά, τα ρομπότ χωρίς οδηγό και ποιος θα πρέπει να έχει υποχρεωτική ασφάλεια. Πώς ορίζεται το ηλεκτρονικό πρόσωπο. Αυτό που έχει σημασία είναι λοιπόν με βάση τον κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς να δούμε πώς θα ορίσουμε την έννοια της ευθύνης μέσα στα πλαίσια της ε, τεχνητής ευθείας Γι' αυτό θα πρέπει να νομοθετήσουμε διαφορετικά επειδή η Ευρώπη ξεπεράστηκε από την επανάσταση της πληροφορικής από τους Αμερικανούς και στον τομέα των μεταφορών με την αποτυχία του Γκαλιλαίου και υπέρ του GPS. Ο κύριος Μάγερ στην έκθεση αυτή προτείνει να ε, υπογραμμιστεί η μείωση ατυχημάτων ε, με βάση τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που θα ισχύει για τα οχήματα, όμως θα πρέπει να υπάρχει και θέμα αστικής ευθύνης στην περίπτωση αυτόματων οχημάτων. Επίσης θα πρέπει η Κομισιόν να δει τις τεχνολογικές εξελίξεις εκ του για να μειωθούν και οι ρηπογόνες εκπομπές. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την αυριανή βιομηχανία με βάση τη συνεργασία κατασκευαστών, δημοσίων αρχών, ερευνητών, καταναλωτών κλπ. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ποιότητα μεταφοράς δεδομένων προς και από τα οχήματα και τις υποδομές για να υπάρχει προστασία της ιδιωτικής ζωής και των οχημάτων. Επίσης, να μην υπάρχει η χνηλάτιση των οχημάτων και να μην μπορεί να γίνει πειρατεία κατά αυτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λουίς Δεκράντες Πασκάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την αντικαταστάτρια του κυρίου ε, Μάιερ. Σίγουρα ζούμε σε μια εποχή τεχνολογικών αλλαγών και επαναστάσεων. Θα πρέπει να δεχτούμε ότι υποκαθίσταται ο άνθρωπος, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων υπέβαλε μία έκθεση επί του θέματος. Ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε τις προάλλες ότι δεν θα θυμάται η ιστορία της πράξης αλλά τα σφάλματά μας και αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να υπάρχουν εγγυήσεις. Μιλάμε για αυτόματα οχήματα και τη ρομποτική, με ατυχήματα βεβαίως, με δυστυχήματα. Και γι' αυτό μας είπε ο κύριος Μάιερ τι πρέπει να προσέξουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αστική ευθύνη, η ευθύνη και η προστασία των δεδομένων. Έχει μεγάλη σημασία να υπάρξει μία κοινοπραξία για τον ορισμό της ευθύνης. Γιατί ο άνθρωπος όταν οδηγεί φέρει ευθύνη και γι' αυτό και συνάπτει και ασφάλεια. Στην περίπτωση της Uber γίνονται και έχουν γίνει προσφυγές σε σχέση με κριτήρια ευθύνης. Γι' αυτό υπάρχει και νομικό κενό. Και μέσα στα πλαίσια της επικουρικότητας οι κοινοπραξίες ε, ασφαλιών ε, μιλάνε για περίπτωση αστικής ευθύνης εκεί όπου πραγματικά υπάρχει ε, ευθύνη και φυσικά θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την απονομή δικαιοσύνης σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα κάνω ορισμένες υποδείξεις και θα υποβάλω και τροπολογίες σε σχέση με την κοινή ευθύνη σε ορισμένες επιμέρους περιπτώσεις. Το θέμα της επικουρικότητας είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για μια νομική βάση της επικουρικότητας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο δικό δίκτυο υπάρχουν και διασυνοριακά ζητήματα. Γιατί γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία για να καλύπτει ε, όλη την ευρωπαϊκή δαφική επικράτη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μάιερ μπορούμε να δεχτούμε την έκθεση αυτή για γνωμοδότηση και θα συνεισφέρουμε με γνωμοδοτήσεις για να συνεισφέρουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά. Ευχαριστώ, Πέτερ Φαντάλεν. Με συγχωρείτε που θα μιλήσω αγγλικά, κύριε Πρόεδρε, αλλά κύριε... Ο κύριος Τουζινόσκη δεν είναι εδώ και μου έδωσε τι παρατηρήσεις του στα αγγλικά. Λοιπόν, ο κύριο Τούζουνόφσκι ευχαριστεί τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότηση, το οποίο θεωρεί μια καλή βάση για την περαιτέρω εργασία. Είναι πεπισμένο πως η τεχνολογική πρόοδο, όπω φαίνεται από την έρευνα και την ανάπτυξη, θα καταφέρει να ανταποκριθεί στι κύριε τεχνολογικές προκλήσει. Όμω, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθούν τα νομικά ζητήματα. Ο του Ζενόφσκι θα ήθελε να κάνει κάποια σχόλια στην ε, γνωμοδότηση και κυρίως θα εστιάσει σε δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα θέλει να τονίσει την κρίσιμη σημασία που έχει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δορυφορικής ε, Πλοήγησης, τα συστήματα Γκαλιλαίο και Έθνος. Επίσης, Υπάρχει μέλλον στα έξυπνα συστήματα μεταφορών, όμως γίνονται έτσι ακόμα πιο δύσκολες οι αυτόματες μεταφορές όσον αφορά την αξιοπιστία των συστήματων δορυφορικής πλοήγησης. Δεύτερον, σωστά ο εισηγητής εστιάζει στα αυτόματα οχήματα. Όμως, ο κύριος Τοζουνόφς και ο σκιώδης εισηγητής μας θα ήθελε να υπενθυμίσει και τους υπόλοιπους τρόπους μεταφορών και θα ήθελε να αναφερθεί συγκεκριμένα στα μη επανδρομένα αεροσκάφη και στην ισορροπημένη έκθεση της κυρίας Φώστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ. Ματέις Φαν Μίλτενμπερκ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθώ στην τελευταία παρατήρηση του κυρίου Φαντάλεν. Φαίνεται πως ε, ακριβώς ε, εδώ πέρα ε, φαίνεται ότι ο καλός ο καπετάνιος ε, στην Φορτούνα φαίνεται. Δικαίως αναφερθήκε ο κύριος Φαντάλεν στα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το θέμα πάει πέρα από αυτά, πέρα από τα αυτοκίνητα που οδηγούνται μόνα του ή τα πλοία που πηγαίνουν μόνα του. Η Rolls αναπτύσσει ήδη σχετικέ τεχνολογίες. Μιλάμε για μετρό, για λεωφορεία που κάνουν δρομολόγια στις πόλεις. Οι μεταφορές λοιπόν τη ρομποτικής είναι πάρα πολλέ ε, στον τομέα των μεταφορών και βεβαίω εδώ πέρα έχει σημασία να ε, λάβουμε υπόψη τους εθνικούς και ευρωπαϊκού κανόνες για την χρήση της ρομποτικής. Η λέξη κλειδί νομίζω είναι εδώ πέρα ο καλύτερος συντονισμός για να καταλήξουμε στη χρήση της ρομποτικής θα πρέπει να προωθηθεί η ασφάλεια και βέβαιως να είμαστε αρκετά ευέλικτοι για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και το τι γίνεται με τα αυτοκίνητα που είναι αυτόνομα και να τα σε μεγάλη κλίμακα. Υπάρχει μια Ολλανδική εταιρεία στο Άμστερνταμ που αναπτύσσει ένα σύστημα το οποίο παρατηρεί ακριβώς τα συστήματα και το οτιδήποτε βλέπει στον δρόμο όλα τα αντικείμενα. Επίσης, τι ζήτημα ιδιωτική ζωής. Και βέβαια το θέμα είναι το τι γίνεται με την μετάδοση των δεδομένων, με την ε, ψηφιακή ασφάλεια και τέλος βεβαίως την ευθύνη σε περίπτωση ατυχημάτων. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να υπάρξει η σωστή ε, χρήση των, αυτοκι... των αυτοματοποιημένων οχημάτων και λοιπόν, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δρέψουμε τους καρπούς αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων εάν ε, έχουμε γρήγορα, ορίσουμε γρήγορα κάποιους κανόνες και αν θέλουμε πραγματικά η Ευρώπη να έχει έναν παγκόσμιο ρόλο σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες και στο πλαίσιο της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων γρήγορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δίτερ Λίμπρη Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ε, τον εισηγητή, παρά το ότι απουσιάζει. Νομίζω ήταν ε, μια καλή αρχή, αλλά δεν πάνε αρκετά μακριά τα πράγματα. Η ρομποτική δεν είναι μόνο αυτόματα οχήματα, αλλά και μη επανδρομένα οχήματα και τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρθηκαν. Αυτόνομα οχήματα οπωσδήποτε θα δώσουν νέα όθηση στις οδικές μεταφορές Οπότε δεν πρέπει να κοιμόμαστε, θα πρέπει η Ευρώπη να ενισχυθεί μέσω της ενίσχυσης του νομικού πλαισίου για την έρευνα, την κατασκευή και τις δοκιμές αυτομάτων οχημάτων. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα ζητήματα ευθύνης δεδομένων ηθικής να προσαρμόσουμε τους νόμους. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Έχω μία σύντομη παρατήρηση. Ήμασταν στην Τσεχία και είδαμε και αυτόματους σιδηροδρόμους. Δεν αφορά μόνο τα, τους δρόμους. Στο Βερολίνο ήδη πριν από 20 χρόνια αυτόματα οχήματα στο μετρό, αλλά δεν το δεχόταν ο κόσμος. Και τελικά υπάρχει κάποιος ε, μπροστά για να δέχεται ο κόσμος να μπει στο τρένο, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτόματα. Πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτό, για να μην επικεντρωνόμαστε, εν πάση περιπτώσει, μόνο στους δρόμους, γιατί και αυτόματα να γίνουν όλα τα αυτοκίνητα, και από ό,τι φαίνεται θα γίνει έτσι, γιατί είχε πει και ο, ο πριν από 44 χρόνια ο Δήμαρχο τότε ο Σοσιαλδημοκράτη του Μονάχου τα αυτοκίνητα δολοφονούν τι πόλει μα και θα πρέπει κάτι να γίνει. Λοιπόν και αυτόματα να γίνουν όλα τα αυτοκίνητα και με ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πάλι θα υπήρχε το πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να τα χρησιμοποιήσουμε στοχευμένα για να σώσουμε τις πόλεις, το κλίμα και τους ανθρώπους Λοιπόν, να δώσω τώρα τον λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στην Επιτροπή σας, στην Επιτροπή Τραν. Καλωσορίσατε, λέει ο Πρόεδρος. Ως προς την έκθεση του κυρίου ε, Μέιερ θα ήθελα να κάνω ορισμένα συμπληρωματικά σχόλια. Σε σχέση με την οδική ασφάλεια καταλαβαίνουμε ότι είχαμε εκθέσει τα τελευταία δύο χρόνια για την οδική ασφάλεια και βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση ατυχημάτων σε αυτό το τομέα, γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις νέες οδούς της ρομποτικής για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να μειώσουμε τα ατυχήματα ε, γιατί το 90% των ατυχημάτων οφείλονται σε ανθρώπινο σφάλμα. Η DG Move, η Γενική Διεύθυνση Move, ε, θέλει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που να διέπει τα FEE ρομπότ e αυτό το master plan είναι και το πρώτο ε, ορόσημο έτσι ώστε να ακολουθηθεί αυτή η ατζέντα της Επιτροπής σε σχέση με το σημείο 3. Ο ο εισηγητής ζητά συνδεσιμότητα μεταξύ συστημάτων και υπό την Ολλανδική ε, προεδρία αυτό είχαμε πει ακριβώς, ότι δηλαδή ε, μαθαίνουμε ε, μέσω ε, βίωσης, μάθησης διαδικασίας μάθησης, εκμάθησης για να έχουμε καλύτερη νομοθεσία από τα θεσμικά όργανα. Με βάση αυτή τη διαδικασία μάθησης σε σχέση με την ασφαλή διάδραση θα θέλαμε να υπάρχει αυτή η συνδεσιμότητα γιατί ε, ε, φανταστείτε τι θα γίνει αν όλα τα οχήματα στην ουσία είναι αυτόματα. Τι θα γίνει. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχουν πάλι συμφορήσεις και θα κάθεται κανείς στις ουρές διαβάζοντας την εφημερίδα του σε σχέση με την ε, ρομποτική και τα θέματα ασφάλειας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και η προστασία προσωπικών δεδομένων, η αναθεώρηση του κανονισμού και συνεργαζόμαστε με εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε να φτάσουμε σε κατευθυντήριες γραμμές που θα μας βοηθήσουν για να υπάρχει προστασία και σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίως ευχαριζόμαστε, ε, ευχόμαστε και σας ε, εξίσου καλή συνεργασία όπως αυτή που ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια με τον συνάδελφό σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, η Μαρίν Κριστίν Νοτού για να δώσει την απάντηση. Κοιτάξτε, θα διαβάσω τα σχόλιά σας στον κύριο Μάγερ από ό,τι καταλαβαίνω θα τον βρουν σύμφωνο. Μιλήσαμε για την ανησυχία νομικής ασφάλειας, επικουρικότητας, απόρριτου των δεδομένων και την επέκταση της ρομποτικής με όλες τις δικλίδες ασφαλείας και βεβαίως θα διαβιβάσω και τα σχόλια της Επιτροπής. Ελπίζω λοιπόν η έκθεσή του να εγκριθεί ε, χωρίς πρόβλημα από το Κοινοβούλιο, την Ολομέλη. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Α, με συγχωρείτε, η προθεσμία καταθέσεις τροπολογιών, βέβαια. 5 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Έχουμε τώρα τα δύο τελευταία θέματα, τα υπαριθμών 10 και 11. Στατιστικές της μεταφοράς εμπορευμάτων στην εσωτερική ναυσιπλοεία και τι στατιστικέ σχετικά με σιδηροδρομικέ μεταφορέ όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτε και ατυχήματα. Ο ένας, ε, για, το, για το πρώτο θέμα ο κ. Μπα Έικχαουτ και για το άλλο είμαι η εισηγητή ο ίδιο. Το αποτέλεσμα των τριμερών διαλόγων ήδη έχει εγκριθεί σε διαφορετικέ ημερομηνίε από την Επιτροπή. Στο μεταξύ, το Συμβούλιο Υπουργών έχει επίση εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση τον συμβιβασμό. Γι' αυτό Πρόκειται απλώς για τυπικό θέμα τώρα η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών, δηλαδή οι τροπολογίες μπορούν να κατατεθούν σε δεύτερη ανάγνωση βέβαια από τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών, όμως θα, θα ε, πάψει να ισχύει ο συμβιβασμό ακόμη και αν μια μόνο τροπολογία εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό ε, η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών ορίζεται 29η Ενάτου ε, μέχρι τις 10. Ε, Βεβαίως, εγώ είμαι πάντοτε υπέρ της ενεργούς, ενεργούς συμμετοχής μας. Ελπίζω αυτή τη φορά, ωστόσο, να μην κατατεθεί καμιά τροπολογία. Όμως, τυπικά είναι δυνατόν αυτό και γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος να κάνω τη σχετική ανακοίνωση. Η κυρία Μάισνερ, εγώ συμφωνώ απολύτως. Είμαι και για τα δύο αυτά θέματα σκιώδη συγγήτρια των φιλελευθέρων. Και πιστεύω ότι πραγματικά έχει φτάσει, έχουμε φτάσει στο συμβασμό, έχει κλείσει ο συμβασμό να μην τον αγγίξουμε. Σε ευχαριστώ για την υποστήριξή σου για ε, τα θέματα των μεταφορών. Δύο χρόνια χρειάστηκε για τα δεδομένα, δηλαδή για τις μεταφορές των σιδηροδρόμων. Γιατί δεν ήθελαν να συμμετάσχουν, δεν ήθελαν να συνεργαστούν οι δύο θεσμοί. Είπα στον ίδιο τον Τίμερμανς ότι δεν μιλούμε για ε, καλύτερη, μιλάμε εδώ για χειρότερη τελικός νομοθεσία. Γι' αυτό συμφώνησαν Ευρωστάτ και ΕΡΑ και μου είπαν μοιάζει εδώ σαν να συνάπτεται η ειρήνη μετά από 30 πόλεμο. Πάντως καλά, καλό ήταν που δείξαμε υπομονή γιατί τώρα είναι και οι δύο πλευρές ικανοποιημένε. Θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε στην Ολομέλεια βεβαίω. Ελπίζω, όπως είπε και η Γιζίνη Μάισνερ, να μην κατατηθεί καμιά τροπολογία. Πολύ καθαρά πράγματα. Ε, λίγη εδώ τώρα η σημερινή συνεδρία και θα συνεχίσουμε τώρα ε, κυκλισμένο των θυρών με τους συντονιστές.